Α Ας ξεκινήσουμε. Ξεκινούμε την επιτροπή μας. Αμέσως μπαίνουμε στην θέση 7 θέση του Κοινοβουλίου για το σχέδιο προπολογισμού του 2011 όπως τοποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Πρέπει να δώσουμε τρεις θέσει. Δίνω αμέσως το λόγο στην κυρία Μακίνες για την ε, παρουσίαση του σχεδίου γνωμόδοτησή της. Και κατόπιν θα προχωρήσουμε στην ε, ψηφοφορία. Μάιναντ, έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη σε αυτό το σημείο, γιατί είναι πολύ σύντομη και ήδη γνωστή στου αδέλφου ω προ το περιεχόμενό τη γνωμοδότηση. Αύριο ψηφίζει η Επιτροπή των Προπολογισμών για το τμήμα το σχετικό με τη γεωργία για τον προπολογισμό και εκεί ίσω πια να χρειαστεί μια συζήτηση για το πώ ε, κρίνουμε την έκβαση αυτή τη προφορία. Τι τροπολογίε, όπω ξέρετε, έχουμε εμεί που προτείνουμε να απορριφθούν. Το περιεχόμενό τους είναι αρκετά σαφές νομίζω και οι συνάδελφοι ελπίζω να ακολουθήσουν τις συστάσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Βολαιότητα. Έχετε όλοι τον κατάλογο ψηφοφορίας. Αν ναι, να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Διανατάσεως των χειρών. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε συνολικά την γνωμοδότηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστούμε τη Μάιρετ. Όπως σας είχα αναγγείλει, προχωρούμε αμέσως στο σημείο 10 της σημερινής διάταξης για να επιτρέψουμε τον συνάδελφο Ταραμπέλα να φύγει νωρίτερα γιατί έχει ορισμένα προβλήματα. Ε, είχαμε εγκρίνει χτες ήδη την αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Το στρατηγικό πλαίσιο της Ένωσης για την παροχή βοήθεια στι αναπτυσσόμενε χώρε ώστε να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει που έχουν να κάνουν με την επισητιστική ασφάλεια. Η Μάιρα Ντεπαυτού ζήτησε το λόγο. Όχι. Έλεγα λοιπόν στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βοήθεια των αναπτυσσόμενων χωρών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της, πρόκληση της πρόκλησης αεπισητιστικής ασφάλειας. Ο, η συντάξη της γνωμοδότησης είναι ο κύριος Ταραμπέλα. Αναλάβαμε να επεξεργαστούμε μια γνωμοδότηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής. Δίδω λοιπόν αμέσω το λόγο στον Μάρκ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τη γνωμοδότηση. Μάρκ, έχει το λόγο. Καταρχάς, πρώτα, ευχαριστώ που αλλάξατε το ράδιο για να μπορέσω να πω και σε άλλη επιτροπή. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση μπορεί να έχει ένα περιορισμένο πολιτικά χαρακτήρα, δεν είναι εξαρτητικό στο μέτρο που θα ήθελε. Γι' αυτό ζητώ εξ αρχής και θα το επαναλάβω στο τέλος της παρέμβασής μου, να μην τροποποιούμε χωρί λόγο τη γνωμοδότηση και μπαίνοντα σε θέματα που δεν είναι γεωργικού χαρακτήρα. Θα εξηγήσω. Στην εισήγησή μου, ωστόσο, θα αναφερθώ σε μερικά σημαντικά ζητήματα που τα αναφέρω παρεπιπτόντω ε, στη γνωμοδότηση. Σε δέκα σημεία και πολύ συνοπτικά να σα πω. Πρώτον, να ευχαριστήσω τι υπηρεσίε τη Γραμματεία τη Επιτροπής, ιδιαίτερα την κυρία Σεύσο Μπέργκερ, που μου έδωσε έξυπνε. Ε, συμβουλές της υπηρεσίας της Επιτροπής ε, για την ανακοίνωση για την επιστημιστική ασφάλεια των αναπτυσσομένων χωρών, ένα θέμα που ασχολείται άμεσα και με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βασική αρχή, αναγκαιότητα να βλάβουμε αμέσω, να λάβουμε τα κράτη-μέλη επίγνωση τη ανάγκη να υπάρξουν νέε επενδύσει, εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων και μείωση των χρεών των πλέον θυγωμένων χωρών. Επίση, να εκμεταλλευτούμε την γνωμοδότηση αυτή για να επιβεβαιώσουμε το δικαίωμα των λαών στη διατροφή η επισητιστική κυριαρχία, ένα θέμα, έναν όρο που τον προτιμώ από τον όρο ασφάλεια, γιατί ασφάλεια σημαίνει η παροχή προϊόντων και η μη, το μη, ο μη βλαπτικό χαρακτήρα των προϊόντων. Ενώ ε, η κυριαρχία σημαίνει ότι κάθε περιοχή του κόσμου, κάθε τμήμα του κόσμου θα μπορεί να έχει επαρκή διατροφή για τους πληθυσμούς της. Η επισητιστική κυριαρχία λοιπόν πρέπει να γνωριστεί και να τύχει υποστήριξη από την Ένωση, κάτι που θα πρέπει να εμφανίζεται σαν βασικό στοιχείο, βασικό δικαίωμα στη διατροφή. Τρίτο σημείο. 70% των ατόμων που υποφέρουν από πείνα στον κόσμο ανήκουν στην Ήπεθρο για να ζουν στην Ήπεθρο. Αυτό απαιτεί ε, την ενίσχυση της, των καλλιεργειών επιβίωσης. Ωστόσο πρέπει να αναπτύξουμε και στρατηγικέ για να ενθαρρύνουμε τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δίνοντας έμφαση στον θεμελιώδη ρόλο των γυναικών και των συνεργατικών δομών μικρών παραγωγών, να ενισχύσουμε την τοπική παραγωγή και να, ε, γενικεύσουμε τις μικρο, τα μικροδάνεια. Επίσης, τέταρτο, πρέπει να υποστηρίξουμε σαν Ένωση τις περιφερειακές συνεργασίες για την ενίσχυση μιας ε, εξοικονόμησης καλλιεργειών. Πέμπτον, απελευθέρωση και κερδοσκοπία στις τιμές πρέπει να καταπολεμηθεί. Χρειάζεται μία ρύθμιση της αγοράς με μία πιο διάφανη αντιμετώπιση της ελευθερίας παραγωγής προς όφελος των μικρών παραγωγών. Έκτον, δεν θα το αναφέρω. Η παραγωγή με βιώσιμο τρόπο και με, μικρό, και με λιγότερο ενεργοβόρο τρόπο θίγει και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επτά, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην, ε, χρήση των γεωργικών προϊόντων ως αγροκαυσίμων. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον ε, η παραγωγή αυτή, αλλά δεν θα πρέπει το ένα να έρχεται σε η παραγωγή γεωργικών προϊόντων να έρχεται σε αντιπαράθεση με την παραγωγή προϊόντων για ενέργεια. 8. Η γη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Πρέπει να προστατεύσουμε τα εμπράγματα δικαιώματα στην γη, ε, δίνοντας δικαίωμα σε όλους να μπορούν να καλλιεργήσουν κάποιο τμήμα γης. 9. Να υπάρξει ένα εκπαιδευτικό και πρόγραμμα και πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιτρέπει στους νέους να συνεχίσουν και να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους να παράγουν, περιορίζοντας την ε, έξοδο από την ύπεθρο και μειώνοντας την φτώχεια. Τέλος, να ενισχύσουμε την έρευνα που χρηματοδοτείται από το δημόσιο στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας. Θα μπορούσα να μπω και στα 9 δισεκατομμύρια τόμου που θα χρειαζόμαστε να να θρέψουμε το 2050 και να έχουμε μια πολιτική ε, γεννήσεων ε, ευρύτερο, την, τις συνέπειες μια σειράς επιδημιών όπως του AIDS που συνεχίζει να πλήττει πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, να καταπολεμηθεί η διαφθορά, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να χτυπήσουμε τη διαφθορά, γι' αυτό επανέρχομαι στο αρχικό μου θέμα. Εάν υποβάλλετε τροπολογίες και θέλω να ακούσω πρώτο όσους θέλουν να μιλήσουν, ιδιαίτερα τους οικειώδεις συγκητές, θα σας ζητούσα να μην κάνετε τροπολογίες που μιλούν για την αύξηση της θερμοκρασίας, για άλλα ζητήματα άσχετα με το δικό μας, γιατί θα βαρύνουμε το κείμενο και θα μειώσουμε τη δύναμη του μηνύματος που θέλουμε να περάσουμε. Ελπίζω να υπάρξει μια πλειοψηφία μαζί μου στην γνωμοδότηση αυτή για να βιώσουμε ότι η γεωργία επιβίωσης και οι περιφερειακές ε, ανταλλαγές είναι αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βάλει μπροστά στις συνεργασίες της με τις ε, ε, αναπτυσσόμενες χώρες να βελτιώσουμε την ε, επισητιστική κυριαρχία των χωρών αυτών και να βοηθήσουμε την επιβίωση των ε, πληθυσμών. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ και Δίνω μέσως το λόγο στους σκιώδεις συγητές. Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την γνωμοδότησή του. Υποστηρίζω όλα τα σχόλια και προσθέτω ακόμη ένα σχετικό με την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν το δεκαετία του 90 κατά 17% αφιερωμένη στην ε, ε, γεωργική ανάπτυξη αναπτυσσόμενες χώρες ενώ το 2008 έπεσε στο 8%. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει εμείς από τη Γεωργική Επιτροπή να υπογραμμίσουμε πως χρειάζεται να επαναδεσμευτούμε στην υποστήριξη της ε, γεωργίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος και εξηγεί και γιατί η μεταφορά τεχνογνωσίας έρευνας και όλα αυτά τα σημαντικά θέματα που συζητήσατε, που αναφέρατε, δεν έχουν προχωρήσει στον αναπτυσσόμενο κόσμο ιδιαίτερα. Πολύ καλή γνωμοδότηση λοιπόν, αλλά νομίζω ότι πρέπει ιδιαίτερα να επισημάνουμε τη συγκεκριμένη πτυχή ως Επιτροπή Αρμόδια για τα θέματα της Γεωργίας. Και χθες εξάλλου συζητήσαμε όλο το θέμα του δικαιώματος σε φαγητό, σε τροφή και πώς μπορούμε αυτό να το υποστηρίξουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε λοιπόν να στηρίξουμε την μικρή κλίμακας ε, γεωργία, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ε, τις λεγόμενες απλής επιβίωσης που ε, είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση των τροφίμων ανά τον κόσμο ε, με ιδιαίτερη έμφαση στην γεωργία στις αναψώμενες χώρες. Η κυρία Γέγκλε έχει το λόγο πρώτα. Χωρίς μικρόφωνο. Το μικρόφωνο της ομιλήτρας είναι κλειστό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαρίστησα τον ε, εισηγητή κύριο Ταραμπέλα και σημείωσα ότι συμφωνώ 100% με τα όσα ε, έχει συμπεριλάβει στη γνωμοδότησή του, όπως και η κυρία Μαγκίνες. Έχουμε ακούσει πολλές επικρίσεις, ιδιαίτερα από τις οργανώσεις των γεωργών, ε, για το ότι είναι λίγα τα χρήματα που πηγαίνουν στην αναταξιακή βοήθεια για την γεωργία, ενώ είναι, πολλά τα, είναι αρκετά υψηλά τα ποσά στους υπόλοιπους τομείς της αναταξιακής βοήθειας. Θα πρέπει λοιπόν ιδιαίτερα να αναφερθούμε στα θέματα της γεωργίας. Πρέπει τα χρήματα, τα κονδύλια που διαθέτουμε να αφιερώνονται ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας. Αυτή είναι η μόνη μου πρόταση πρόταση, κατεπίγουσα πρόταση, δεν καταβάλω ιδιαίτερη τροπολογία γι' αυτό, αλλά δεύτερο θα ήθελα να πω και είναι πολύ σημαντικό και επίγον ότι ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω και εκείνοι που ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να το επισημάνουν, ε, να ε, μεριμνήσουμε να είναι σύμφωνες και συντονισμένες με τις δικές μας επιλογές οι κυβερνήσεις. Εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν πόλεμοι, ε, ταραχές, δεινά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες, να προσφέρουμε χειραβοηθείας, αλλά χρειαζόμαστε τη σύμπραξη και των κυβερνήσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο χωρίς απαραίτητα να καταθέσουμε τροπολογία θεωρώ σημαντικό και θα πρέπει να μπει στο κείμενο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μάρτιν Χέσλιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική έκθεση και για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη που είναι, αφήνει μάλλον μια πικρή γεύση για να το πω κομψά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορθώς το ανάστημα και να αναλάβει μόνη της τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πείνας και φτώχειας. Ο Μάρκο Ταραμπέλα αναφέρεται ιδιαίτερα στους ε, γεωργούς, στους ε, καλλιεργητές με κρίση κλίμακας ε, στις χώρες του τρίτου κόσμου, στις τρίτες χώρες μάλλον. Είναι ιδιαίτερος ο λόγος νομίζω για τον οποίο θα πρέπει να στοχεύσουμε στους ανθρώπους αυτούς. Το έχουμε επισημάνει και σε εκθέσεις πριν από δύο χρόνια σε μια έκθεσή μας ότι δηλαδή οι επιστηστικές ανάγκες ανά τον κόσμο μπορούν να επιληθούν εάν να δώσουμε στήριξη στους γεωργούς αυτούς των τρίτων κρατών, ταυτόχρονα όμως των απτυσσομένων κρατών, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει και να ε, τους στηρίξουμε ως προς τα δικαιώματά τους. Επίσης ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι πού πηγαίνουν οι πόροι, αλλά και ε, οι, πόροι με κάθε έννοια και ενεργειακοί δηλαδή πόροι. Μίλησε επίσης ο κύριος Σταραμπέλα για διαδικασίες οι οποίες ε, μπορεί να οδηγούν εφόσον ε, συνεχίσουμε τις εισαγωγές ε, αλκοόλης σε στρέβλωση των συνθήκων της αγοράς και πάντως σε δυσμενείς συνέπειες για τους γεωργούς των τρίτων αυτών κρατών, των αντισωμένων κρατών και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα το κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσουμε την προαγωγή τέτοιου είδους εισαγωγών. Εν τέλει και συνολικά νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε μέσα από τη γνωμοδότηση αυτή την ευθύνη που έχουμε έναντι των χωρών του τρίτου κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντέση έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τα όσα υπόθηκαν ήδη. Ο Μάρκ Ταραμπέλα είναι ικανός συνάδελφος, βρίσκεται σε καλά χέρια η γνωμοδότηση. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνει πολύ καλή έκθεση, πολύ καλή γνωμοδότηση. Τελευταίες εβδομάδες και μέχρι και τελευταία Κυριακή είχα πολλές επαφές ε, με εκπροσώπους γεωργών και από την Αφρική, γενικά οργανώσεις ε, μικρών ε, εκμεταλλεύσεων και έμαθα πράγματα τα οποία με έχουν συγκλονίσει όπως παραδείγματι το γεγονός ότι στο Κονγκό, στην Αφρική αλλά όχι μόνο στο Κονγκό οι Κινέζοι έχουν αγοράσει 2,8 εκατομμύρια εκτάρια γεωργική γη και όχι μόνο στο Κονγκό αλλά σε πολλές άλλες αφρικανικές χώρες και δεν είναι μόνο οι Κινέζοι αλλά και πολλοί άλλοι και πολλές ήταν οι αφρικανικές οργανώσεις γεωργών οι, οποίοι μου κρούν τον, οι οποίες μου κρούν τον κόντρα του κινδύνου ότι ε, πρέπει εμείς οι Ευρωπαίοι να αντιδράσουμε. Φοβούνται ότι θα χάσουν από τα χέρια τους και τη γη τους την ίδια και ότι θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί, κυρίως στις μικρές εκμεταλλεύσεις στην Αφρική, εάν πωλείται η γη κατά αυτόν τον τρόπο. Και επίσης η αναπτυξιακή βοήθεια που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η σχετική αναπτυξιακή πολιτική στην Αφρική αντιμετωπίζει πολλές επικρίσεις και λέγεται ότι δεν είναι ε, στοχευμένη σωστά. Πρέπει λοιπόν να ανασταθμίσουμε αυτή την αναπτυξιακή βοήθεια και να τη στοχεύσουμε κατά τρόπον ώστε πράγματι να αποβαίνει εις όφελος των ε, ανθρώπων της περιοχής, εκείνων που έχουν πραγματική ανάγκη και να μην επιτρέψουμε στους Κινέζους με την ε, παρέμβαση τους αυτή στην γεωργία στην Αφρική να προξενήσουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες. Ο κύριος Γιάννη, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς τον συνάδελφο Ταραμπέλα για την έκθεσή του. Θα πρέπει η έκθεση να μας επιτρέψει μια ευρύτερη θεώρηση της αναπτυξιακής πολιτικής μέσα από τη γεωργία. Θα ήθελα δύο-τρεις λέξεις μόνο να πω με την ελπίδα ότι θα μπορέσει ο συνάδελφος Ταραμπέλα να τις εντάξει τις ιδέες μου μέσα στο κείμενό του. Πείνα λοιπόν και καταπολέμηση της πείνας δεν, είναι μόνο, δεν βρίσκει τη λύση της μόνο μέσα από παροχές αρρωγής και βοήθειας. Χρειάζονται δημοκρατικές και σταθερές σχέσεις στα αναπτυσσόμενα κράτη. Χρειάζεται καταπολέμηση της διαφθοράς. Η απουσία διαφθοράς είναι μια από τις ελάχιστες προϋποθέσεις Αυτό ισχύει φυσικά και για τη γεωργία, γιατί δεν μπορεί να είναι ασφαλής ο γεωργός στην ε, ε, ε, καλλιέργεια της γης του, εάν οι συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας δεν υφίστανται. Και δεύτερο, χωρίς να θέλουμε βέβαια να ευλογάμε τα γένια μας, οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ειδωτήσεις των εξαγωγών που έχουν σαν στόχο την ε, ε, στήριξη ορισμένων ε, προϊόντων θα πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα να μην πλήττονται τα τρίτα κράτη, τα κράτη του τρίτου κόσμου και η μικρότερη αυτή παραγωγή. Και τρίτον, νομίζω θα πρέπει ιδιαίτερα να φροντίσουμε με τα μέτρα που θα εισάγουμε ή μη τι άλλο να μην βοηθούμε τους λεγόμενους κακούς, αυτούς δηλαδή οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ήδη πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, και επίσης, συμπληρώνω, θα πρέπει να έχουμε και το θάρρος κονδύλια τα οποία διαθέτουμε για την αναπτυξιακή βοήθεια να τα ελέγχουμε ε, ως προς το πώς και πού αξιοποιούνται. Εδώ δεν μιλάω μόνο για τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι δαπάνες της αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να επαληθεύεται πού πηγαίνουν γιατί έστω και εκ των υστέρων τα σφάλματα που έχουν επαχθεί θα πρέπει να τα διορθώνουμε γιατί μπορούμε να τα διορθώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ή δυνατόν να ενσωματωθούν αυτές οι ιδέες στο κείμενό σας. Χάσφορτ παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ κατά Μάρκ για την έκθεση του. Θα συμφωνήσω με τα περισσότερα από τα σχόλια του. Εδώ το γενικότερο πλαίσιο μας δείχνει ότι ο παγκόσμιος πληθυσμό θα συνεχίσει να αυξάνεται και βλέπουμε τις συνέπειες της φτώχειας ε, στον πλανήτη. Όταν κάποιοι ξεφεύγουν από την φτώχεια βλέπουμε να οδεύουν ε, προς μια διατροφή δυτικού τύπου ε, υψηλή, υψηλά ποσοστά κατανάλωσης πρωτενη, πράγμα που αποτελεί αποτίμαλων και καλλιέργειε, μεγάλε εκτάσει γης, απασχολεί και τη βιομηχανία καυσίμων που χρειάζεται την ε, συνδρομή από την ζάχαρη, τα, το καλαμπόκι, τα σιτηρά. Όλα αυτά λοιπόν θέτουν τους φτωχότερους ανθρώπους του πλανήτη σε ιδιαίτερα μενεκτική θέση και οι αρνητικές συνέπειες για αυτούς είναι ιδιαίτερα δυσανάλογες. Γι' αυτό ο ΟΗΕ ε, δημοσίευσε μια προειδοποίηση για την επιστηστική ασφάλεια και είπε ότι εάν δεν αυξηθεί η παραγωγή τροφίμων μέχρι το 2030, με την αύξηση του πληθυσμού θα υπάρχει σοβαρή επιστημιστική κρίση. Υπάρχει λοιπόν ε, επιτακτική ανάγκη ηθικού χαρακτήρα ε, για τι αναπτυγμένε χώρε, ιδίω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναλάβουν δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερο εισαγωγέα τροφίμων. Εισάγουμε το ισοδύναμο 35 εκατομμυρίων εκταρίων ε, τροφίμων κάθε χρόνο, το μέγεθος της Γερμανίας. Η παγκόσμια αγορά για να επιτρέψει την εισαγωγή τέτοιων ποσοτήτων τροφίμων οδηγείται ουσιαστικά σε αύξηση των βασικών αγαθών, των τιμών των βασικών αγαθών. Και επαναλαμβάνω εδώ ότι είμαστε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας παγκοσμίω σε τρόφιμα. Συνεισφέρουμε δηλαδή στις, στην αύξηση των τιμών των βασικών αγαθών και ουσιαστικά στερούμε από τους φτωχότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να μπορούν να τραφούν τελικά. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη για μας, ηθική ανάγκη, και πραγματικά θέλω αυτό το μήνυμα να περάσει, να είναι ηχηρό, ε, είναι επιτακτική ανάγκη τα ανεπτυγμένα κράτη, ιδίω η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναλάβουν ε, τι ευθύνε του. Ε, προκειμένου να επεκτείνουμε την παραγωγή μα και να καλύψουμε τι δικέ μα τι ανάγκε, τη δική μα τη ζήτηση, αλλά πρέπει να έχουμε και μηχανισμού που να λειτουργούν, ώστε να μην είναι βλαβερέ οι συνέπειε τη δική μα ανάπτυξη για τον αντισώμενο κόσμο και τη δική του γεωργία. Ευχαριστούμε κύριε Χάσπορθ. Ο κύριο Σιλβέστρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι σκληρός εισηγητής για το ΕΛΚ για την ε, έκθεση αυτή και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ταραμπέλα. Θα προσυπογράψω στο σύνολο της παρέμβασής του. Όμως, ενώ η Επιτροπή μας συζητά για την ε, σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τι συμβολή μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προ τι αναπτυσσόμενε χώρε και την επιστημιστική του ασφάλεια, μιλάμε για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Θα πρέπει λοιπόν η τοποθέτησή μα να έχει μια διαφορετική βαρύτητα και έχει και ιδιαίτερη σημασία. Θα ήθελα να επικεντρωθώ εδώ στην ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει τα ερχόμενα χρόνια στον διπλασιασμό τη παραγωγή τροφίμων για να καλύψει τι ανάγκε του παγκόσμιου πληθυσμού που θα αυξηθεί κατά 3,5 δισεκατομμύρια άτομα μέχρι το 2050. Πρέπει λοιπόν να παράγουμε περισσότερο, καλύτερα και με τρόπο πάντοτε πιο βιώσιμο τέσσερα τουλάχιστον στοιχεία έχουν οδηγήσει σε τέσσερα ε, έχουν οδηγήσει στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης. Η επέκταση των μη επεξεργασμένων τροφίμων, η αύξηση των αναγκών, η παραγωγή των ε, βιοκαυσίμων και εδώ στέκομαι μόνο στο 7ο σημείο από τα 10 που απαρίθμησε ο συνάδελφο Ταραμπέλα και εδώ θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο και να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Είναι κομβικό το σημείο αυτό. Και έπειτα και η επιρροή των κλιματικών αλλαγών που επηρέασαν την ε, σοδιά και καθίστησαν, καθίστησαν ακόμη πιο δύσκολη την καλλιέργεια συγκεκριμένων προϊόντων. Κατά την άποψή μου λοιπόν υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην νομοδότηση αφού ούτω ή άλλω συμφωνούμε στην προσέγγιση μα και δεν θέλουμε να την επιβαρύνουμε ιδιαίτερα με πάρα πολλέ τροπολογίε θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλεία για τα προϊόντα, για τα τρόφιμα πρώτη ανάγκη, αλλά να φροντίσουμε και για τι αναπτυσσόμενε χώρε που δεν μπορούν να αντισταθούν στι συνέπειε τη επιστημιστική κρίση και τι δυσκολίε τη αγορά. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για να αυξήσουμε την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφέ, τι ζωοτροφέ και αυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καυσίμων. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τι παραδοσιακέ καλλιέργειε. Οφείλουμε επίση να έχουμε εντατικότερη γεωργική καλή δραστηριότητα προκειμένου να περιοριστούν οι τιμέ και αύξηση τους για του καταναλωτέ, αλλά να επιτρέψουμε και μεγαλύτερο κέρδο για του γεωργού καθώ και οικονομική ανάπτυξη. Επίση να πρέπει να επιτρέψουμε τις, ε, την ανταλλαγή καλών γεωργικών πρακτικών όπω επισημαίνει και ο συνάδελφο Ταραμπέλα για να διευκολύνουμε την ανάπτυξη και τη διοργάνωση φορολογικών συστημάτων όριμων ε, στο πλαίσιο της ε, καλής γνώσης των γεωργικών πρακτικών και προκειμένου να είμαστε και αυτάρκης από ενεργειακής άποψης. Εδώ θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο σημείο αυτό, γιατί θεωρώ ότι η ενεργειακή αυτάρκεια μέσω των γεωργικών συστημάτων, των συστημάτων γεωργικής παραγωγής, είναι ένα ε, σημείο καθοριστικό. Θα μπορούσε αυτό να απαλλάξει τους, τους μηχανισμούς γεωργικής ε, παραγωγής από τις διακυμάνσεις των τιμών στον τομέα της ενέργειας. Εδώ η Ευρώπη δεν είναι ακόμα αρκετά αυτόνομη και αυτάρκης. Επίσης, τα προϊόντα ενέργειας ε, με δεύτερης γενιάς, ε, με τη χρήση γεωργικών προϊόντων, όπως το βιοδίζελ από αραβόσιτο, οδηγεί σε αλλαγή της τιμή του ραβοσίτου. Αυτό είναι σίγουρα ένα πλεονέκτημα από την άποψη της ενέργειας, αλλά είναι σίγουρα επίσης ένα πρόβλημα ως προς την επισητιστική προμήθεια ραβοσίτου. Εδώ μιλάμε λοιπόν για προϊόντα χίδιν, τα οποία θα πρέπει να τα προκρίνουμε στην παραγωγή τους. Έτσι λοιπόν μπορούμε να σκεφτούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον πυρήνα των ε, ε συγκεκριμένων γεωργικών προϊόντων, τον, τον, τα κουκούτσια της ελιάς λόγου χάρη, τα περισεβούμενα προϊόντα, τα υπολείμματά τους και εκεί να τα αξιοποιήσουμε. Κάποιες φορές επίσης πρέπει να προωθήσουμε τις βιολογικές καλλιέργειες, κάτι που είναι ευκταίο για την Ευρώπη, αλλά εδώ χρειάζεται ανάλογη προσπάθεια για να μην ξεπεράσουμε την παραγωγή των παραδοσιακών καλλιεργιών. Χθε ε, στην Επιτροπή μα συζητήσαμε το θέμα αυτό και ο συνάδελφο Ντε πάντοτε σημειώνει την σημασία τη συμμετοχή των γυναικών στι γεωργικέ δραστηριότητε. Για την παρουσία λοιπόν των γυναικών στο γεωργικό τομέα είναι σημαντικό να συζητήσουμε περαιτέρω στην Επιτροπή μας. Υπάρχουν εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την παρουσία των γυναικών στον γεωργικό πληθυσμό. Μιλάμε για ομάδες ε, ευάλωτες των γυναικών καθώς και εθνικές μειονότητες. Ε, πιστεύω ότι με τον συνάδελφο Ταραμπέλα θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε από κοινού τροπολογίες με ένα πνεύμα ε, συνεργασίας. Ευχαριστούμε κύριε Σιλβέστρης. Ο κύριος Καπόλα Σάντος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά δεν μπορώ να παραλείψω να εκφράσω την άποψη της ομάδας των σοσιαλιστών, την εκτίμησή μας δηλαδή, για το έργο, για τη δουλειά του συναδέλφου Ταραμπέλα και ένα θέμα τόσο επίκαιρο. Ήθελα λοιπόν να εκφράσω δημοσίως την στήριξη της ομάδας μας για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ η Αντιπρόεδρος κυρία Πότς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ προς τον εισηγητή. Υπάρχουν δύο ή τρία ενδεχόμενα μεγάλα προβλήματα στο πλαίσιο αυτό. Πρώτον, κάτι που ανέφερε ο κύριος Ντες. Η εξαγορά τεράστιων εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης σε φτωχές χώρες που τώρα είναι ακαλλιέργητες αλλά που μπορεί να μπορέσουν να γίνουν ε, πολύ πιο αποδοτικές αργότερα. Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα την Αφρική. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Ο πλούσιος κόσμος έχει την ικανότητα να πληρώσει έχουμε τη βούληση να πληρώσουμε ώστε να βάζουμε στο αυτοκίνητό μας βενζίνη από εθανόλη που την παίρνουμε από το στόμα των φτωχών ανθρώπων στις φτωχές χώρες. Δεν θα έπρεπε να κατασκευάζουμε καύσιμα αυτοκινήτων από τρόφιμα. Υπάρχουν πολλά προϊόντα στη γεωργία και στην δασοπονία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για βιοκαύσιμα, όχι ωστόσο τρόφιμα. Τρίτο θέμα που αφορά πάλι την Αφρική. Η έλλειψη δομών απόδειξης της κυριότητας της αγροτικής γης. Ποιος έχει την χρήση, την ε, κυριότητα της γης οι γυναίκες, οι φτωχοί καλλιεργητές έχουν ιδιοκτησιακές, ε, ε, έχουν ιδιοκτησίες. Μπορούμε να δημιουργήσουμε σε κοινωνίες, στις κοινωνίες αυτές τους θεσμούς που θα είναι αναγκαίοι για να διατηρηθεί το κράτος δικαίου και μια σειρά βασικών ελευθεριών Στι χώρε αυτέ. Ευχαριστώ κύριε Πόλσον. Η κυρία Κλάση έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή η εκθέση, αλλά ταυτόχρονα και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να καλέσω τον συνάδελφο Ταραμπέλα να αξιοποιήσει την ευκαιρία που μας προσφέρεται να προσδιορίσουμε τι θέλουμε εμείς ε, να κάνουμε για την ε, επιστηστική ασφάλεια και για μια ασφαλή επιστηστική κατάσταση στα αναπτυσσόμενα κράτη. Αυτό που δεν μπορώ να αντιληφθώ και που διαρκώς μου προξενεί πολύ ανησυχία και δυσκολία είναι το γιατί θα πρέπει σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στον ολόκληρο τον κόσμο να βρίζουμε ένα τον άλλον. Αυτό που έχουμε να κάνουμε μόνο είναι να συνεργαστούμε και να κάνουμε μια καλή δουλειά. Γιατί θα πρέπει πάντοτε να θέτουμε το δάκτυλο από τον τύπο των ήλων δεν πρέπει να γνωρίζουμε καλύτερα τι πράττει η αριστερά και τι πράττει η δεξιά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς είναι δυνατόν στην ανάπτυξη παραδείγματι να μιλούμε για ε, την ε, μάλλον να μην συζητούμε καν την διάθεση της υπερβολικής, η παραγωγής μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη αυτά. Α, όταν έρχεται όμω συζήτηση, η Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη μου λέει: Κοιτάξτε, εμεί δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι είναι θέμα τη Γενική ε, Διεύθυνση τη Γεωργία να αναλάβει τη σχετική απόφαση. Ε, λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να θέσουμε το δάκτυλο από τον τύπο των ήλων, να πούμε ότι δεν υπάρχει επαρκή συνεργασία μεταξύ των δικών μα των ε, υπηρεσιών και ότι πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε να έχουμε μια ουσιαστική και καλή προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βόλσκι, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πιστεύω ότι πρέπει να επανεξετάσουμε την ευρύτερη πολιτική στον τομέα της γεωργίας της Ένωσης. Ε, αναφέρθηκε ήδη ότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή σημαντικά μέχρι το 2010. Αναφέρθηκε και το πρόβλημα της εξαγοράς αγροτικών γεών στην Αφρική. Οι Ινδίοι και οι Κινέζοι αγοράζουν εκεί γη γιατί έχουν μεγαλύτερη ε, φαντασία από εμά. Λέμε τώρα ότι την εξουσία την έχουν αυτοί που έχουν το πετρέλαιο. Αυτό θα αλλάξει στο μέλλον. Αυτός που θα έχει την ισχύ θα είναι αυτός που έχει τη γη. Θα είναι ακριβή η παραγωγή τροφίμων και όποιος έχει τη γη θα μπορέσει να ελέγχει το εμπόριο. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε γιατί ακόμα ζούμε στην εποχή ε, του περιορισμού της ε, γεωργικής παραγωγής και της αποσύνδεσης της ε, παραγωγής με την γη. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον εν ώψη προκλήσεων όπως της έλλειψης τροφίμων που θα γίνει ένα στρατηγικό αγαθό. Θα πρέπει να πληρώνουμε για το αγαθό αυτό. Δεν πληρώνουμε τώρα. Ε, είμαστε, το είπε και κάποιος άλλος, η μεγαλύτερη εισαγωγή τροφίμων και θα συνεχίσουμε να είμαστε να αλλάξουμε πολιτική. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο Άλμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ να διευκρινίσω κάτι σε σχέση με τα όσα είπα νωρίτερα. Αυτό που είπα νωρίτερα για τους Κινέζους που έχουν αγοράσει 2,8 εκατομμύρια εκτάρια στο Κονγκό, προφανώς δεν το κάνουν γιατί θέλουν να καλλιεργήσουν τρόφιμα για τους Αφρικανούς που ζουν στην περιοχή, αλλά γιατί θέλουν να παράγουν, παράγουν προϊόντα τα οποία θα εξάγουν μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει περίπου ένα εκατομμύριο Κινέζων στην Αφρικανική Ήπειρο ήδη εγκατεστημένων εκεί που φυσικά επηρεάζει πάρα πολύ τα δεδομένα μια τέτοια ε, έντονη παρουσία. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν που έχουν να κάνουν με την Αφρική θα πρέπει να τα κοιτάξουμε με πολύ μεγάλη προσοχή γιατί έχουν και εσωτερικές ρίζες πολλές φορές. Στη Ζιμπάμπου επί παραδείγματι όταν υπάρχουν επαρκείς πόροι ε, φυσική, όταν η γη παράγει αρκετά, πώ είναι δυνατόν να πεινάει ο κόσμο. Και όμω ολόκληρε περιοχέ Ζιμπαμπού πεθαίναν από, το, από την πείνα πριν από μερικά χρόνια. Στη Ζάμπια είδαμε το ίδιο. 27 γεωπόνους έστειλε στο εξωτερικό η κυβέρνηση της Ζάμπιας ε, για να μπορέσουν να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερη απόδοση της γης τους. Αυτό τι λέει, λέει ότι δεν χρειάζεται μόνο χρήματα να ρίχνουμε για να βοηθούμε τους ανθρώπους αυτούς, αρκεί να μάθουν μόνοι τους να βρίσκουν τις λύσεις για τα προβλήματά τους. Αυτό όμως προϋπόθεση απαρέκλητη έχει μια σταθερή διακυβέρνηση, σταθερές κυβερνήσεις στα αφρικανικά κράτη. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το, το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, κύριο Βιμ Όλτοφ, ζητώ από τον κύριο Ταραμπέλα, θέλει να απαντήσει ή όχι. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, σημειώνω όλες τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Και βεβαίω με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρατηρώ ότι η γενική τάση της έκθεσης βρίσκει του περισσότερου σύμφωνους. Πάντω, θα είμαι πολύ προσεκτικό για τι τροπολογίε που θα υποβληθούν, για αρχέ που είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιώσουμε εκ νέου. Πράγματα που ίσω δεν είπα στην πρώτη μου παρέμβαση, αλλά άκουσα κάποια σχόλια, όπω αυτά του κυρίου Γιάρ. Ε, Κάποια τα έχω ήδη συμπεριλάβει, είχα σκοπό να τα συμπεριλάβω, θα τα συζητήσουμε, δεν τα είπα όλα στα προκαταρτικά μου σχόλια. Ε, φαντάζομαι ότι οι σκιώδεις εισηγητές και ο κύριος Σιλβέστρης του ΕΛΚ, δεν ξέρω τα ονόματα όλων των ε, συναδέλφων που θα είναι σκιώδε εισηγητές, αλλά θα συναντηθούμε σίγουρα και θα συζητήσουμε τροπολογίες, συμβαστικέ λύσεις, ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε την ίδια βούληση να επιβεβαιώσουμε την ε, βασική κυριαρχία που θα πρέπει να έχει η γεωργία για σκοπούς ε, διαβίωσης και κάλυψη πρώτων αναγκών και την προστασία του γεωργικού κόσμου. Ε, εδώ όταν μιλάμε για ελάφρυνση του βάρου των δανείων, αυτό σίγουρα θα πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με την επένδυση σε πολιτικές που θα βοηθούν, θα διευκολύνουν τη ζωή των ε, πληθυσμών και δεν θα λειτουργούν εναντίον τους. Ευχαριστούμε Μάρκ. Ο, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο κ. Σόλτοφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή σας για την πολύ καλή επισκόπηση δέκα σημαντικών σημείων που προκύπτουν από την ανακοίνωσή μας. Η ανακοίνωση αυτή αφορά την ε, ένδια, την πείνα σε παγκόσμιο επίπεδο το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας. Περίπου 100 εκατομμύρια ακόμη άνθρωποι δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε ε, τρόφιμα. Το θέμα είναι λοιπόν πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διευκολύνει τι αναπτυσσόμενε χώρε να έχουν πρόσβαση. Η ανακοίνωση δίνει μια ιδιαίτερη προτεραιότητα στις γεωργούς των μικρών εκμεταλλεύσεων και καλλιεργιών. Αυτό το μήνυμα έχει περάσει πολύ σωστά και στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα όμως να επισημάνω κάποια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα η ανακοίνωση αυτή συνοδεύτηκε και από μια ακόμη ανακοίνωση από συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ για την επισητιστική βοήθεια, συνδρομή όταν υπάρχουν λοιπόν κατεπίγουσε καταστάσει με προβλήματα πείνα, κάποια ιδιαίτερη κρίση, ε, υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που συμπεριλαμβάνει και προτείνει αυτή η ανακοίνωση. Το γεγονό ότι δημοσιεύτηκαν αυτέ οι ανακοινώσει ταυτόχρονα οφείλεται στο γεγονό ότι κάποιε φορέ στην Επιτροπή το δεξί και το αριστερό χέρι και συναντιούνται και το έναν ή διτάλο και τα δυο το πρόσωπο. Εδώ λοιπόν μιλάμε για θέματα πείνας και για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το αρνητικό φαινόμενο. Η συζήτησή σα πολύ σωστά στάθηκε σε ένα από τα σημεία που αφορούν τι αναπτυσσόμενε χώρε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η κατοχή γη, τα προγράμματα ιδιοκτησία γη. Η ανακοίνωση τη Επιτροπή ε, ε, υποδεικνύει μια σειρά από τρόπου που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στην Αφρική ιδιαίτερως, διότι η γη δεν είναι το μόνο πρόβλημα εκεί. Το άλλο πρόβλημα είναι η πρόσβαση σε πόρους. Δηλαδή, η γη και το νερό είναι πράγματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν παράλληλα. Και φαντάζομαι ότι και η συζήτηση του Κοινοβουλίου θα το λάβει υπόψη το στοιχείο αυτό. Αυτά σε ό,τι αφορά της ενθερμόντες δράσεις μου στην όλη συζήτηση που έγινε εδώ. Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά να δώσουμε διευκρινήσεις και από τη δική μας πλευρά προς τον εισηγητή, προκειμένου να τον διευκολύνουμε. Σας εύχομαι πάντως ε, με ιδιαίτερη σύνεση να καταλήξετε στα τελικά σας συμπεράσματα στην έκθεση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Και σε αυτό το σημείο, Μάρκ σου Είμαστε στα χέρια σου για την επεξεργασία του σχεδίου έκθεση και στην επόμενη συνεδρίασή μα θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του γερμανικού μονοπωλίου αλκοόλης. Εφόσον είμαι συγκητής, μου δίνω το λόγο και πολύ γρήγορα να σας παρουσιάσω την έκθεση. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά την συζήτηση που είχαμε για το γερμανικό μονοπόλιο αλκοόλης στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας και επειδή είναι συγκητής για το θέμα αυτό, υπέβαλε ένα σχέδιο γνωμοδότησης που επί τη ουσίας αντικατοπτρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ορισμένε βοήθειες προς την Γερμανία στον τομέα της παραγωγής αλκοόλης ως το 2017. Είχαμε από κοινού με άλλους συναδέλφους εκφράσει κάποιους ενδιασμούς ιδίως ό,τι αφορά την παράταση της παρέκκλησης μετά την ημερομηνία του 2013 όταν θα ισχύει πλέον μια νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ωστόσο, μετά τις διαβεβαιώσεις των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεδομένων των περιορισμένων διαστάσεων και την σημασία για την οικονομία της υπαίθρου των αποστακτηρίων που λαμβάνουν τις βοήθειες, θεωρώ ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις αρχικές μας αμφιβολίες. Μπορούμε λοιπόν την παρέκκληση όπως την προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη δεχτούμε. Η μόνη τροπολογία που υπέβαλα σκοπό έχει να αυξήσει τη διαφάνεια και τον δημοκρατικό έλεγχο στο όλο σύστημα, ζητώντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβιβάζει στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την ετήσια έκθεση της Γερμανίας για την σταδιακή μείωση του μονοπωλίου, τον περιορισμό του μονοπωλίου. Θα κλείσω ε, ευχαριστώντας την κυρία Γιαγκλέ, η οποία διοργάνωσε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την εβδομάδα του Στρασβούργου, επιτρέποντάς μας να γνωρίσουμε τα μικρά αποστακτήρια του μέλλον δρυμού ε, στη Γερμανία. Και είδαμε τι σημασία έχουν αυτού του είδους οι μικρές επιχειρήσεις για την οικονομία της ε, περιοχής αυτής. Με αυτά τα προκαταρτικά λοιπόν σχόλια ανοίγω την συζήτηση και έπειτα θα δώσω το λόγο και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Γιάγκλη, έχετε ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε και θέλω να ευχαριστώ θερμά και για την γνωμοδότησή σας αλλά και για την αιτιολόγηση. Έχουμε νομίζω μια πολύ καλή περιγραφή της κατάστασης και πιστεύω ότι αυτή τη ε, διαφοροποίηση στην οποία προβαίνεται την ε, συζητούν και στη Γερμανία. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει στην ε, Γερμανία μετά το 2017 αλλά είναι ένα πρόβλημα πάνω απ' όλα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Εμείς θα πρέπει να βρούμε ως κράτος τη λύση. Είναι σαφές νομίζω το ποιος είναι ο τρόπος να ξεφύγουμε να καταργήσουμε ε, αυτό το μονοπόλιο είναι δεδομένο και μετά την επίσκεψη στο Μέρα να ότι ο δρόμος αυτός δεν γυρίζει πίσω, είναι μονόδρομος. Χαίρομαι για το ότι μέσα στην έκθεση προβλέπεται η ετήσια ενημέρωση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ε, υπόθεση αυτή του μονοπωλίου και παρακαλώ τους συναδέλφους ε, την έκθεση να την ε, εγκρίνουν με τις τροπολογίες που έχει τώρα, να μην καταθέσουν περισσότερες τροπολογίες οι οποίες ενδεχομένω να ανέτρεπαν το κείμενο και να οδηγούσαν και εμάς και τον ε, εισηγητή βέβαια στην ε, αναγκαστική διαπραγμάτευση μέσα από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Η βάση την οποία έχουμε νομίζω είναι καλή, την έχουμε συζητήσει και διαπραγματευτεί και υπογραμμίζω για άλλη μια φορά ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από τον γερμανικό κορβανά και όχι από τον ευρωπαϊκό. Κάτι που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν οι συνάδελφοι είναι ότι τα προϊόντα αυτά μόνο στη Γερμανία μπορούν να απολυθούν. Τα προϊόντα αλκοόλης δεν έχουν δηλαδή σχέση ανταγωνιστική με άλλα αντίστοιχα προϊόντα που πολλούνται σε κράτη-μέλη όπως η Γαλλία, η Αυστρία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο μέσα στη Γερμανία μπορούν να απολυθούν. Και έτσι θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει καν κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Παρακαλώ λοιπόν να εγκρίνετε την έκθεση ω έχει με τι τροπολογίε του εισηγητού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριο Ρόντουστ. Η κυρία Ρόντουστ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ υποστηρίζω την, ε, το σχέδιο εκθέσεως ε, του Παόλου για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την εκπνοή του γερμανικού μονοπωλίου αλκοόλης για το 2010 που, αρχι... που όπως οριστεί αρχικά θα προκαλούσε βέβαια πολλές δυσκολίες στους μικρούς κυρίως παραγωγούς. Ε, όπως είδαμε και από τις επισκέψεις μας επί τη ευκαιρία της εβδομάδας στο Στρασβούργο, ε, είναι αυτή η παραγωγή αλκοόλης ο τρόπος επιβίωσης για αρκετές από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και έτσι μια πρωτοβουλία από την κοινή γεωργική πολιτική που θα μπορούσε να μας επιτρέψει το 2013 να έχουμε μια πολυλειτουργική και βιώσιμη αλλά και εκτεταμένη ε, επιβίωση αυτών των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, μικρότερες δηλαδή και ε, μικρότερε γεωργικέ εκμεταλλεύσει οι οποίε θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν και τη διαφύλαξη αρκετών θέσεων εργασία. Εδώ μπορούμε, πιστεύω, και με στη βιοπικιλότητα να συμβάλλουμε, αλλά και στη διαφύλαξη των παραδοσιακών δομών και τρόπων εργασία ε, στην ύπεθρό μα και τεράστιο Μέλλον Δρυμό. Η συζήτηση για το μονοπόλιο, για την αλκοόλη, είναι νομίζω γνωστή, όπως είπε και η Ελίζα Μπεθιέκλε. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο ε, έχει επιπτώσει τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, αλλά μόνο στο γερμανικό. Και όπως υπόθηκε, και εγώ χαιρετίζω την πρόταση. Λυπούμε μόνο για το γεγονός ότι τα προϊόντα δεν είναι δυνατόν να απολυθούν εκτός της Γερμανίας. Το λέω αυτό ε, μόνο χαριετιζόμενοι, γιατί απλώς όταν τα προϊόντα αυτά είναι τόσο νόστιμα που θα άξιζε τον κόπο να μπορεί ο καθένα και από τη Γερμανία να τα γευθεί. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη προ τι μικρότερε επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ο Μάλτιν. Ευχαριστώ. Ναι, ήταν όντω πολύ ωραία η επίσκεψη στον Μέλλον Αδρυμό προσπαθώ να μην παρασυρθώ από το πάθος και από τους ε, ατμούς της αλκοόλης. Εν πάση περιπτώσει ένα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα. Είναι κάτι το οποίο έχει την ιστορία του και νομίζω είναι σαφές και για όσους γνωρίζουν την κατάσταση και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που είναι στην περιοχή και ασχολούνται με την παραγωγή αυτή ότι του μένουν ακόμα έξι χρόνια. Μια παράταση μόνο, τίποτα άλλο. Μετά τελειώνει αυτή η ιστορία του μονοπωλίου. Ιδιαίτερα θα ήθελα να επισημάνω και να χαιρετήσω το γεγονό ότι από την πρόταση βλέπουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ αυτών τα οποία ανέφερε και η κυρία Γιάνγκλη βέβαια, των μικρών επιχειρήσεων δηλαδή, των μικρών αποστακτηρίων συνεταιρισμών αποκαλλιεργειών που συμβάλλουν και στη διαφύλαξη, στη Βάδη Βιτεμπέργη, την ΕΣΥ, τη Βαβαρία ε, της παραδοσιακής γεωργίας και ε, των παραδοσιακών επαγγελμάτων της υπαίθρου που έχουν να κάνουν με γεώμηλα και σιτηρά κυρίως τα αποστακτήριά τους. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα ότι έχουμε να κάνουμε και με επιχειρήσεις οι οποίες σε μια μεταβατική περίοδο ίσως θα είναι σε θέση να αναζητήσουν νέες δυνατότητες ε, διάθεσης των προϊόντων τους, νέες δραστηριότητες ενδεχομένως. Αυτό τον αέρα θα τους προσφέρει η παράταση της ε, περίοδου του μονοπωλίου. Αυτό μπορούμε να τους προσφέρουμε εμείς και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει ένα σαφές μήνυμα με την παράταση Ύστερα από την περίοδο αυτή όμως των έξι ετών που δίνουμε περιθώριο θα τελειώσει η ιστορία του μονοπωλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστώ. Μάρτιν, ο Herbert Hoffman έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα την ανάλυση σας για το πρόβλημα. Να προσθέσω ωστόσο δύο λόγια για αυτό που είπε ο κ. Χόισλινγκ. Η επίσκεψη που διεξάγαμε μας έκανε νομίζω να καταλάβουμε καλά ότι το σχέδιο αυτό είναι χρήσιμο για να μην μπει σε κίνδυνο ολόκληρη η δομή που δημιουργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή αυτή ε, και που έχει σημασία για την περιοχή αυτή. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η δομή αυτή, ως έχει τώρα, πάνω από 100 παραγωγούς και ε, πολιτές σε ένα χωριό, δεν είναι βιώσιμη Ούτε τώρα, ούτε το 2017. Άρα είναι αναγκαίο να υπάρξει μία δέσμευση και της εθνικής κυβέρνησης και της τοπικής κυβέρνησης για βελτίωση των δομών. Η... Το κόστος, θα υπάρχει μία ε, ε, ε, βραδία έξοδος, θα έχει κέρδη για τα lender που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακριβώς για να αλλάξουν τη δομή πωλήσεως των προϊόντων αυτών που είναι εξαιρετικά και που πιστεύω ότι είναι κρίμα. Δεν χρειάζεται να έχουμε μονοπόλιο σε αυτά τα προϊόντα υψηλή ποιότητα. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν το κράτος να χρησιμοποιήσει τα λίγα χρόνια που έχει μπροστά του μαζί με τους παραγωγούς και τις ενώσεις παραγωγών ώστε να δημιουργήσει ένα σύστημα πωλήσεων που δεν θα είναι τόσο τοπικοποιημένο αλλά ε, εκτενέστερο επιτρέποντας τα εξαιρετικά αυτά προϊόντα να βρουν μια πραγματική αγορά. Πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση για τους ε, παραγωγούς ε, μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ, Χέρμπερτ. Ο κύριος Βατσεβόφσκι, αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ θα υπερψηφίσω την έκθεση διότι καταρχάς, καταρχήν μάλλον υποστηρίζω τις μικρές επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τους μικρούς αυτούς επιχειρηματίες. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ενεργή εμπλοκή των Γερμανών συναδέλφων η διατήρηση της παραγωγής αυτής μπορεί να μείνει στη Γερμανία. Δεν θα συμφωνούσα ωστόσο ότι ε, αποτελεί στρέβλωση των αγορών. Παρότι λέμε ότι η πώληση πρέπει να γίνεται μόνο στη Γερμανία, ε, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η γερμανική αγορά είναι τμήμα της ευρωπαϊκής. Ένα κομμάτι λοιπόν της ευρωπαϊκής αγοράς θα έχει κορισμό από το προϊόντα αυτού, αυτά. Οπότε η παραγωγοί, οι αλκοόλης δεν μπορούν, από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν μπορούν να να πωλήσουν εκεί. Είναι παγκόσμια η παραγωγή. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον πρόεδρο ή τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Γιατί αυτή η εξαίρεση, ποια είναι η, πηγή, η πηγή ε, της εξαίρεσης αυτής για τους γερμανούς παραγωγούς. Μόνο το ότι μπαίνει στη μέση γερμανική κυβέρνηση και στην Πολωνία έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Ξέρω πολλά από στα κτίρια στην Πολωνία, στην περιοχή μου, που παράγουν αλκοόλια από αραβόσιτο, ζουν, πουλάνε, χωρίς ενισχύσεις. Θα μπορούσαν λοιπόν να συνεχίσουν την παραγωγή τους. Ε, μήπως λοιπόν η γερμανική κυβέρνηση απλώς έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από άλλες. Άκουσα τα επιχειρήματα πάντως και είμαι πεπισμένος ότι η παραγωγή είναι καλή, αλλά η εξαίρεση είναι που δεν μου αρέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Ο George Line. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ από την πλευρά των φιλελευθέρων να πω ότι στηρίζουμε την έκθεση του κ. Ντακάστρο. Αντικατοπτρίζεται και κάποια θέματα όπως τα συζητήσαμε εδώ στην Επιτροπή μας και σαφώς μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει σοβαρή επίδραση στην ευρωπαϊκή αγορά από την στήριξη αυτών των προϊόντων ε, αφορά τη γερμανική αγορά. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκή θα μπορούσε να μας πει αν υπάρχει δυσανάλογος αντίκτυπος ή όχι. Πάντως, η γερμανική κυβέρνηση προσπάθησε να στηρίξει αυτά τα μικρά αποστακτήρια Να στηρίξει λοιπόν αυτά τα μικρά αποστακτήρια προκειμένου να προσαρμοστούν στην σταδιακή μείωση τη κρατική ενίσχυση, νομίζω ότι είναι ορθή. Δηλαδή θα πρέπει να την προβλέψουμε αυτή τη μεταβατική περίοδο και να υπάρξει παράταση όπω προτείνει και δέχεται η έκθεση. Ευχαριστούμε, Τζόρτζ. Κύριο ε, Ευχαριστώ. Στη συνάντησή μας χθες... Στη συνάντησή μας χθες με τον Επίτροπο Τσόλος μίλησα για, μιλήσαμε για τη διαφοροποίηση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας όπου χρειάζονται διαφορετικά εργαλεία και μέσα στήριξης. Ε, σας είχα πει χθες ότι ανησυχώ ιδιαιτερός για το μέλλον της ΚΑΠ διότι Υπάρχει υπερβολική τάση προς απλούστευση και ενοποίηση του όλου συστήματος. Εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα πρέπει να υπάρξουν διαφορετικά μέτρα στήριξη, διαφορετικά εργαλεία, προκειμένου να διατηρήσουμε θέσεις εργασίας και την παρουσία προϊόντων σε μικρές τοπικές αγορές. Είμαι λοιπόν ε, θερμά υπέρ της ε, συνέχειας, της παράτασης της στήριξης προς τα προϊόντα αυτά. Τα επιχειρήματά μας είναι και πολύ σαφή. Απλώς έχουμε μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ανάλογες καταστάσεις, παρόμοιες καταστάσεις άλλων χωρών θα ληφθούν υπόψη. Πώς τα κατηγοριοποιεί αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς πότε θεωρείται μια εκμετάλλευση μικρής κλίμακας και πότε ένας μικρός παραγωγός φτάνει τα όρια του μεγάλου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριο Ντέσου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αναφέρθηκαν κάποια σημεία από τους αδέλφους που ήθελα και εγώ να αναφέρω. Ε, δεν θα μακρηγορήσω λοιπόν, απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πάολο αλλά και την Ελίζαμπετ που συνέβαλε πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Πάνω απ' όλα πρέπει νομίζω να σημειώσουμε ότι δεν προσπαθούμε να διαφυλάξουμε αυτές τις επιχειρήσεις, να τις ενισχύσουμε, απλώς να τις βοηθήσουμε μόνο να περάσουν από τη δύσκολη περίοδο της προσαρμογής στις νέες συνθήκες μετά τη λήξη του μονοπωλίου. Ούτε νομίζω ότι πρόκειται να πάνε ε, μαζικά ε, ξένοι να αγοράζουν τέτοιου είδους προϊόντα αλκοόλης από τη Γερμανία παρότι είναι τόσο νόστιμα βέβαια όπως υπόθηκε τόσο καλής ποιότητας Όπω είπε και η συνάδελφος νωρίτερα, δεν επιτρέπεται να απολυθούν στο εξωτερικό αυτά προϊόντα, αλλά από την άλλη αυτό δεν μπορεί να σημαίνει ότι μα απαγορεύεται να τα δορίζουμε στο εξωτερικό. Δεν μπορεί ούτε η Επιτροπή να μα απαγορέψει κάτι τέτοιο. Νομίζω λοιπόν αγαπητοί συνάδελφε Ρόντου, ότι μπορούμε να φέρνουμε ο καθένα μα από ένα μπουκάλι ή δύο για να κερνάμε του φίλου μα καμιά φορά. Και νομίζω ότι με την ευκαιρία αυτή ε, υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά ότι επιτρέπουμε στις μικρές αυτές επιχειρήσεις, στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να διαχειριστούν καλύτερα την μετάβαση στην περίοδο μετά, το μετά την κατάρριξη του μονοπωλίου. Άλλωστε πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είναι και η πρώτη φορά, ούτε η μοναδική φορά που εισάγονται παρεκκλήσεις μέσα στη γεωργική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό παρακαλώ συναδέλφους να μας βοηθήσουν να υποστηρίξουν την πρόταση. Ευχαριστούμε, Άλμπερτ. Να κλείσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Νταντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, να ευχαριστήσω την συνάδελφο, την κυρία Γέγκλε, που διοργάνωσε την επίσκεψη τη περασμένη εβδομάδα. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όχι μόνο και για το θέμα που μα απασχολεί, αλλά επειδή μα επέτρεψε να δούμε και κάποια άλλα στοιχεία. Τώρα, προκειμένου, να πω ότι πρέπει να παραμείνουμε στα εξή. Το σύστημα αυτό επέτρεπε σε μικρού γεωργού να έχουν ένα συμπλήρωμα για το εισόδημά του, αρκετά συμφέρον και να παραμείνουν ε, στη θέση του. Είναι λίγε εκμεταλλεύσει έτσι κι αλλιώ στην γεωργική περιοχή που επισκεφθήκαμε. Και χωρί αυτή τη διέξοδο θα είναι, αλλάξει η γεωργική παραγωγή, οπότε θα επηρεαστεί και το τοπίο τη Γερμανία γενικότερα. Αυτά λοιπόν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πρέπει να έχουμε συνέστηση των ε, εξέλιξεων που μπορούν να προκύψουν. Σήμερα μιλάμε για βιοπικιλότητα. Το να καταργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα μακροπρόθεσμα οδηγεί σε ισοπαίδωση ε, του τοπίου, του σκηνικού σε αυτό το μέρο τη Γερμανία. Και κατά τη διάρκεια τη μέρα, όσο υπήρχε το φω του ήλιου δηλαδή, μπορέσαμε να διακρίνουμε το τι κάνουν οι γερμανικές εκμεταλλεύσεις για να είναι εξοπλισμένες με... και να παίρνουν ενέργεια από τον ήλιο με ηλιακές, με ηλιακές γεννήτριες. Εδώ μπορεί βεβαίως να, αν αλλάξει παραγωγή και αντικαταστήσει την παραγωγή αλκοόλης, μπορεί να αλλάξει και αυτή η τροφοδότηση. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πολύ καλά το θέμα αυτό και σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και με το πώς αναζητούν πόρους οι γεωργοί. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς όλους για τις παρεμβάσεις σας και την υποστήριξη στην έκθεση. Να καθησυχάσω και κάποιους συναδέλφους για την ανησυχία που εξέφρασαν Το λέει και η έκθεση, το λέει και η Επιτροπή. Αιτιολογείται επαρκώς η παρέκκληση. Όπως και σε κάθε παρέκκληση ε, προκύπτουν ορισμένα στοιχεία στρέβλωσης. Αυτό είναι αυτονόητο. Νομίζω ωστόσο ότι ταυτόχρονα υπογραμμίστηκε και ο περιορισμένος βαθμός της παρέμβασης, ιδίω η παρέμβαση μόνο από, ότι επιβαρύνει μόνο την ε, Γερμανία, ότι η πώληση αφορά μόνο το γερμανικό έδαφος, και τα προβλήματα ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσουν οι περιοχές αυτές σε περίπτωση που δεν με παρέμβουμε δίνουν απαντήσει. Να υπογραμμίσω επίσης ότι σήμερα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ειδική επιτροπή Γεωργίας, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό, ο κ. Ούιμπερξ προεδρεύων είναι ε, της Βελικής Προεδρίας είναι παρόν και ξεκινά, πρέπει να το υπογραμμίσω αυτό, μια σημαντική δράση κατά εφαρμογή της διεργασίας της Λισαβόνας συνεργασίας των δύο δομών. Ευχαριστώ λοιπόν τον εκπρόσωπο της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας, την εκπρόσωπο της ε, Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας και θα δώσω αμέσως το λόγο αν το ζητηθεί, αλλά να ρωτήσω την Επιτροπή πρώτα μήπως θέλει να μιλήσει. Ε, θέλει να μιλήσει ο εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής. Παρακαλώ. Δύο λόγια μόνο για να απαντήσω σε δύο ερωτήματα τη επιτροπή. Καταρχά, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. για την έκθεση που προτίμασε. Κάποιος ρώτησε από πού προέρχονται, γιατί υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Όπως ξέρετε το γερμανικό μονοπόλιο θεσπίστηκε το 1918. Παρατάθηκε και άλλαξε κατά τη διάρκεια των ετών, αλλά είναι παρέκκληση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για πολύ καιρό. Τώρα θέλουμε να πάψει οριστικά αυτή η παρέκκληση από τις κρατικές ενισχύσεις. Τούτο θα γίνει σε έξι χρόνια. Ένα άλλο ερώτημα αφορούσε το κατά πόσον υπάρχουν μικρά αποστακτήρια σε άλλες χώρες. Βεβαίως υπάρχουν αλλά δεν βρήκαμε αντίστοιχα προγράμματα με αυτά της Γερμανίας σε άλλη χώρα της Ένωσης που να έχει τους κανόνες αυτούς ε, ή τις παρεκκλήσεις από τις κρατικές ενισχύσεις. Άρα θεωρούμε ότι με τον κανονισμό αυτό το 2017 δεν θα υπάρχει πλέον καμία παρέμβαση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων σε κανένα κράτος της Ένωσης. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο ε, ο πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας να του δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Κατέγραψα την ε, συνολική επιδοκιμασία της Επιτροπής σας για την πρόταση αυτή. Φαντάζομαι, όπως διαπιστώνω, ότι θα εγκρίνετε την πρόταση και ελπίζω σύντομα να ολοκληρωθεί η συζήτηση και στο Συμβούλιο. Ωραία λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ όλους, προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Στο σημείο 9 ειδικότερα. Ευρωπαϊκές στατιστικές για τις μόνιμες καλλιέργειες. Η κυρία Νεντέλτσεβα είναι η συγγήτρια. Το ξέρουμε το θέμα. Ξέρουμε την, την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις εκτάσεις, για τις στατιστικές δεδομένα των ε, ε, μονίμων καλλιεργειών. Μαρία, σου δίνει το λόγο για να μας παρουσιάσει την πρότασή σου. Η κυρία, η κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω θα ξεκινήσω με την αιτιολόγηση και μετά αφού πρόκειται και για ανταλλαγή απόψεων θα ήθελα να σας διατυπώσω πολλές από, τις, από τους προβληματισμούς μου, τις απορίες μου, τα ερωτηματικά μου και βεβαίως Περιμένω να ακούσω αντίστοιχα και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων έτσι ώστε με βάση την πρόταση της Επιτροπής ε, να έχουμε ένα κείμενο δικό μας το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των συναδέλφων ε, της Επιτροπής μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπενθυμίσουμε ότι η παραγωγή οπορολαχανικών αποτελεί ε, μία από τις κυρίες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την πρόταση αυτή προσπαθούμε να επικαιροποιήσουμε το υφιστάμενο πλαίσιο, το ισχύον πλαίσιο για τις στατιστικές, αντικαθιστώντας τα δύο ισχύοντα νομοθετήματα από ένα μόνο. Τα δύο ισχύοντα νομοθετήματα, σας πενθυμίζω, είναι ο κανονισμός του 69, 30, 57 και η 109 οδηγία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να επαναλάβω τα επιχειρήματα υπέρ μια επικαιροποίηση, μια ενημέρωση των μαθημάτων, τον τρόπο με τον οποίο πάνω απ' όλα συντάσσονται αυτέ, καταρτίζονται αυτέ οι στατιστικέ είναι αιτήματα τα οποία δεν τυπώνουν εδώ και χρόνια τα κράτη-μέλη αλλά και όλε οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όντω προβλέπουν μια σειρά από τροποποιήσει ε, των νομικών στοιχείων των, στατιστικών, ε, των μονίμων στατιστικών και θα υπενθυμίσω ότι μετά την θέση εφαρμογή των υφεσταμένων νομοθετημάτων έχουν αλλάξει και οι συνθήκε τη κοινή γεωργική πολιτική και η κατάσταση στην γεωργική αγορά εν γέννη έχει σημαντικά μεταβληθεί και ως εκ τούτου η υφιστάμενη πρόταση στόχο έχει να απλουστεύσει τις μεταβλητές και τις έννοιες και να απλουστεύσει σημαντικά τις στατιστικές για τις μόνιμες καλλιέργειες προς όφελος και των χρηστών τους με κατάργηση των, των ετήσιων στατιστικών για τις σπορές και για την πολύ λεπτομερή, υπερβολικά λεπτομερή ταξινόμηση, μάλλον το ευρύ φάσμα στον ίνο. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε έτσι καλύτερες, ε, καλύτερα στοιχεία και πληροφορίες στους χρήστες. Η δε προσθήκη νέων μεταβλητών άλλων ε, ταξινομήσεων αντιστοιχεί βεβαίως στην εξέλιξη της ισχύουσας νομοθεσίας. Για δε πρόσθετες ε, προϋποθέσεις ή απαιτήσει μας λέγεται στο κείμενο, γιατί αυτό ήταν κάτι που με προβλημάτισε και εμένα, ότι στόχος ήταν να μειωθεί ο γενικότερος φόρτος και η γενικότερη στρατιστική επιβάρυνση. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω σε τούτου το εξή ερώτημα προς την Επιτροπή μας. Μιλούμε σε όλο το κείμενο για μια απλούστευση, δηλαδή περιορισμό του ε, φόρτου και για τον παραγωγό, που μας ενδιαφέρει φυσικά περισσότερο, αλλά και για τις εθνικές και ευρωπαϊκές διοικητικές αρχές. Θα ήθελα να παρακαλέσω σε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει περισσότερα στοιχεία να μας δώσει και λεπτομέρειες για αυτή την απλούστευση. Δεύτερον, για την περίοδο κατά την οποία τα κράτη μπορούν να έχουν στη θέση τους για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, στις νέες προϋποθέσεις. Θα ήθελα να διατυπώσω ε, άλλο ένα ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν προβλέπεται καμία περίοδος ε, για προσαρμογή των κρατών μελών σε μία, στις νέες αυτές προϋποθέσεις. Φαίνεται όμως από ό,τι μαθαίνουμε ότι η Γερμανία σκοπεύει να ζητήσει για τα οποροφόρα δέντρα μία ε, περίοδο μετα... Ε, αναπροσαρμογής, περίοδο η οποία από ό,τι φαίνεται δεν θα δημιουργήσει τέτοιες δυσκολίες. Οι Γερμανοί είναι σε θέση να δώσουν τα στοιχεία του είναι έτοιμοι δηλαδή για το 2010 με βάση νέα, την παλαιά οδηγία και ρωτώ εάν υπάρχουν και άλλα κράτη τα οποία έχουν τα δεδομένα αυτά έτοιμα. Και ίσω θα ήταν σκόπιμο, ρωτώ του συναδέλφου, να δώσουν τη γνώμη του, ε, να δώσουμε μια μεταβατική περίοδο για την προσαρμογή αυτή. Και επίση, δεδομένου ότι πρόκειται για μια νομική βάση, μια έκθεση την οποία μα υποβάλλουν προ εξέταση μετά τη θέση ισχύ τη ε, συνθήκη Λισαβόνα. Θα ήθελα να επισημάνω το παράρτημα υπαριθμών 1 και το κείμενο στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι εφόσον πρόκειται για μη ουσιώδη στοιχεία και θα, θα μπορούσαν αυτά να ε, υπαχθούν σε μια διαδικασία εκχωρήσεως εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σχετικό νομοθέτημα. Μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε ε, ότι ε, αυτή η αυτό ο κατάλογο του παραρτήματο 1 μπορεί να ισχύει κατά αυτόν τον τρόπο και ρωτώ του συναδέλφου εάν τα άρθρα 10, 11, 12 τα σχετικά με την εκχώρηση εξουσιών στην Επιτροπή, τι προθεσμίε για την αντίδραση και γενικά τι ε, προνομίε και τι εξουσίε του Κοινοβουλίου μα του βρίσκουν σύμφωνου. Ερωτώ εάν αυτή για να κλείνω η μεταβατική περίοδο μπορεί να ισχύει για τον κατάλογο του παραρτήματο υπαριθμών 1. Αυτό για να ξεκινήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Νεντέλσεβα. Θέλει κάποιος το λόγο, θέλει να ζητήσει κάποιος περισσότερες πληροφορίες μετά από αυτή τη συνθητική παρουσίαση της συγγήτριας που ανοίγει μια σειρά προοπτικών. Θα ζητήσω από την Επιτροπή να απαντήσει. Ο κ. Καρντόσο. Θέλετε να απαντήσετε σε ερωτήσει που έφυγε η κυρία Νεντέλτσεβα. Είναι... Ευχαριστώ. Ξεκινώ ευχαριστώντα την κυρία Νεντέλτσεβα για την πλήρη ολοκληρωμένη εισαγωγή της που περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της πρότασης και της αιτιολόγησής της. στις απαντήσεις θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ζητήματα που έθεσε η κυρία Νεντέλτσεβα. Ε, ζητήματα που φαντάζομαι ότι και πολλοί άλλοι μεταξύ ημών ε, ε, συμμερίζονται. Όπως υπογράμμισε η κυρία Νεντέλτσεβα, η πρόταση αυτή έχει στόχο να αντικαταστήσει κείμενα της δεκαετίας, νομοθετικά κείμενα της δεκαετίας του 70 που άλλαξαν πολλές φορές, αλλά που χρειάζονταν ε, μία βαθιά αναμόρφωση. Γι' αυτό το λόγο, στο πλαίσιο αυτής της ε, στο πλαίσιο της νομοθετικής απλοποίησης και των προσπαθειών μας ε, να μειώσουμε στο μέτρο του δυνατού την επιβάρυνση των αγροτών που δίνουν τις απαντήσεις, παρουσιάζουμε αυτό το νέο κείμενο. Ποιες είναι οι βασικές απλοποιήσεις που εισήχθησαν στο κείμενο. Καταρχάς, υπάρχει το ότι πλέον ζητάμε στατιστικά στοιχεία και δεν κάνουμε έρευνες. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το κράτος μέλος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλες πηγές πληροφόρησης από πέραν των ερευνών. Αυτό θα έχει συνέπειες τόσο σε αυτούς που παρέχουν τις απαντήσεις, τους γεωργούς δηλαδή, διότι ε, ε, εάν η πληροφορία είναι ήδη διαθέσιμη σε άλλα διοικητικά αρχεία δεν χρειάζεται να ζητηθούν εκ νέου. Υπάρχουν αλλαγέ στο, συν, στο, στον αριθμό των πληροφοριών που ζητούνται. Αυτή τη στιγμή ζητούνται στατιστικές για τα πέντε χρόνια για, πέντε χρόνια για τα οποροφόρα, δέκα για τα αμπέλια και κάθε χρόνο για αμπέλια εάν έχει γίνει αλλαγή ε, ε, έκτασης με διαφοροποίηση, αναπεριφέρεια, απόδοση κλπ. Είναι λοιπόν πολλές πλήρεις πληροφορίες που απαιτούνται κάθε χρόνο. Ε, οι πληροφορίες αυτές δεν θα ζητούνται πλέον. Πέραν της μείωσης των απαιτήσεων στοιχείων, βάλαμε και κάποια κατόφλια. κάτω από τα οποία δεν θα χρειάζεται να δίδονται πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα. Άρα δεν καθιστούμε υποχρεωτική την παροχή στοιχείων για μικρές, ε, πολύ μικρές ε, ε, εκμεταλλεύσει κάτω από ένα δέκατο του εκταρίου ή περιοχές όπου η παραγωγή είναι χαμηλότερη από 500 εκτάρια συνολικά. Έτσι φεύγει από τα στατιστικά ένα μεγάλο τμήμα παραγωγών που είναι αυτοί που καθιστούν ε, δαπανηρότερη την πιθανή διεξαγωγή ερευνών ή παραγωγή στατιστικών δεδομένων. Μειώσαμε τις ποικιλίε από 88 σε 18 για τα μήλα, από 64 σε 11 για τις αχλαδιές, από 164 για τα ροδάκινα σε 18. Αν θέλετε μπορείς να τον πλήρη κατάλογο. Μειώσαμε τις τάξεις επικνότητας, τις τάξεις ε, της κλάσης ηλικία, την περιφερειακή κατανομή ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερες περιφέρειες. Υπογραμμίζω τη σημασία των ε, στοιχείων, ε, των περιφερειακών στοιχείων ηλικίε για την καλύτερη κατανόηση των πεθεριών και όλων των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της ε, υπαίθρου. Όλα αυτά απλοποίησαν τα αποτελέσματα, μείωσαν κατά πολύ το κόστος των ερευνών όποτε χρειαστεί να γίνουν τέτοιες έρευνες απογραφής. Για τα στατιστικά δεδομένα των αμπελιών προβλέπουμε όλα τα στοιχεία που ζητούνται να είναι διαθέσιμα στο αμπελοϊνικό μητρό. Να μην χρειάζεται δηλαδή να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες που ζητούνται μπορεί να αντιληθούν απευθείας από τα αρχεία αυτά. Με λίγα λόγια. Αυτές ήταν οι κύριες απλοποίησεις. Σε ό,τι αφορά τη μεταβατική περίοδο, Πιστεύω ότι θα υπάρχει δυνατότητα να εξεταστεί το ζήτημα αυτό και αργότερα. Πρέπει να σας πω ότι ο στόχος ε, της απλοποίησης ήταν να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές χωρίς να προβαίνουν σε δύσκολη και επίπονη δραστηριότητα όπως το παρελθόν, αλλά με πολύ πιο γρήγορο τρόπο. τρόπο. Καταλαβαίνουμε ωστόσο ότι σε κάποιες χώρες ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων γίνεται πολύ νωρίτερα. Οπότε οι προθεσμίες ε, για την πρόταση αυτή που έπρεπε να γίνει νωρίτερα, να συζητηθεί νωρίτερα και να εγκριθεί ελπίζω νωρίτερα, θα μπορεί να αποτελέσουν στοιχείο δυσκολίας για κάποιες χώρες. Ίσως λοιπόν όπως και για αντίστοιχα άλλα νομοθετικά κείμενα να, βρεθεί, να χρειαστεί να βρεθεί συμβαστική λύση. Τώρα για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις Βρισκόμαστε σε μία περίοδο υλοποίηση της νέας συνθήκης. Άρα, έγινε όλο το προπα... ενώ έγινε όλο το προπαρασκευαστικό έργο στο πλαίσιο της παλιάς συνθήκης και με το Συμβούλιο, ομάδα στατιστικών δεδομένων όπου είχαμε ήδη μια πρώτη συνάντηση και όπου τέθηκε το ζήτημα αυτό. Η Επιτροπή λοιπόν βρίσκεται στο στάδιο όπου προσπαθεί να ακούσει τις απόψεις όλων προσπαθώντας να βρει την καλύτερη δυνατή λύση ούτως ώστε να απαντήσει στις θεμητές προσδοκίες των ε, νομοθετικών ε, οργάνων. Δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το δικαίωμα παρακολούθησης. Πρέπει ωστόσο κατά την άποψή μας, να διατηρήσουμε μία ισορροπία μεταξύ των διαδικασιών αυτών που ενδεχομένως μερικές φορές είναι επίπονες και των ε, πιθανών αναγκών προσαρμογής καθώς και της εμπειρίας και των αλλαγών που η εμπειρία θα καταστήσει μάλλον αναγκαίες. Στο παρελθόν πιστεύω ότι η Επιτροπή πάντα έδειξε πως ε, επιθυμούσε να συνεργάζεται στενά με το Κοινοβούλιο για τα κράτη-μέλη για να αποδείξει ότι επιδιώκει τον συντονισμό και θέλει να ακούσει τις προσδοκίες όλων. Πιστεύω λοιπόν ότι και τους επόμενους μήνες και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και της ε, διαμόρφωσης ενός ε, συμβιβασμού που θα εφαρμοστεί κατά πάση πιθανότητα όχι μόνο σε αυτόν τον κανονισμό αλλά και σε άλλους, θα έχουμε την ευκαιρία να βρούμε μία λύση που θα σέβεται τις προσδοκίες όλων. Τελειώνω Να πω δύο λόγια για τη σπουδαιότητα αυτών των πληροφοριών. Η παραγωγή οποροφόρων και αμπελιών είναι σημαντική. Σε τοπικό επίπεδο κυρίως σε ορισμένες περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν μεγάλη πηγή για ένα κομμάτι της υπαίθρου που δεν έχει εναλλακτικέ λύσεις. Ό,τι λοιπόν επιτρέπει να έχουμε καλύτερη γνώση και κατανόηση των στοιχείων αυτών των καλλιεργιών είναι σημαντικό. Ο στόχος είναι η Επιτροπή και οι διάφορες υπηρεσίες της να πετύχουμε αυτό το στόχο. Να έχουμε δηλαδή ταυτόχρονα ένα απλό, ευέλικτο σύστημα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διαφόρων εμπλεκόμενων φορών. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Θέλετε να παρέμβετε, κύριε Ντέλτσεβα. Α, α, συγγνώμη. Κύριος Ντές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων στη συνάδελφο Λεντέλτζοβα, η οποία μπόρεσε να επεξεργαστεί αυτό το τόσο άκομψο θέμα, τις στατιστικές, με αποτέλεσμα στο μέλλον να μην χρειάζεται περιτές στατιστικές, περιτά στατιστικά στοιχεία να καταγράφονται. Από τα όσα άκουσα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω μία ελπίδα ότι μπορούμε να, είναι και, να είμαστε και κάπως πιο αξιόπιστοι στις στατιστικές που έχουμε. Γιατί εδώ και αρκετά χρόνια οφείλω να πω ότι δεν τολμάω να ανοίξω το στόμα μου σε θέματα κατάργησης της γραφειοκρατίας και περιορισμού της γραφειοκρατίας όταν μιλώ με τους εμπλεκόμενους επισκέψεις μου στις διάφορες χώρες διότι το αποτέλεσμα που βλέπω εγώ είναι όχι κατάργηση γραφειοκρατίας αλλά μάλλον ενίσχυση της γραφειοκρατίας και ίσω θα μπορούσαμε εν γέννη να αναπτύξουμε αυτές τις προσπάθειες για κατάργηση της γραφειοκρατίας. Παρακαλώ όλους εμπλεκόμενους να ξεκαθαρίζουν, να απαλλάσσουν τις στατιστικές μας από κάθε περιττό στοιχείο. Πράγμα το οποίο θα σημάνει ως μεγάλο κέρδος την ενίσχυση της αξιοπιστίας των στατιστικών αυτών. Και έτσι μπορούμε, πιστεύω, να περιορίσουμε την περιττή γραφειοκρατία και σε επίπεδο επιτροπής. Ευχαριστώ κύριο Ντόρφμαν έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μπορώ να είμαι πολύ σύντομος, καθώς μπορώ και εγώ να συμφωνήσω προς το περιεχόμενο πλήρως με τα όσα είπε ο κύριος ε, Ντες. Είναι πολύ σημαντικό να καταργήσουμε, να αποδιαρθρώσουμε την περιττή γραφειοκρατία και θα ήθελα να εισαγάγω μία λεπτομέρεια ακόμα ότι το ζήτημα των ε, ορίων, ε, των προσδορισμών, ταξινομήσεων ή των τρόπων μέτρησης δεν είναι ο μόνος, η μόνη λύση στην περίπτωση αυτή. Είναι μια συζήτηση την οποία έχουμε κάνει κατά καιρού. Δηλαδή τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές το καθένα μεθόδους ε, και για λόγους παραδοσιακούς ακόμη για τον υπολογισμό ε, των εκτάσεων Φερρυπίν. Μια έκταση την υπολογίζουν από το η ρίζα ενό δέντρου μέχρι τη ρίζα ενό άλλου δέντρου ή υπολογίζουν ε, Φερρυπίν το εξωτερικό δέντρο μια ε, έκταση μέχρι το επόμενο εξωτερικό δέντρο. Αυτές είναι παραδοσιακές μέθοδοι τις οποίες δεν μπορούμε εμείς να ανατρέψουμε. Πρέπει να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να τις διατηρήσουν εφόσον αποδεδειγμένα είναι ικανοποιητικές χωρίς να επιβαρύνουμε με περιττή γραφειοκρατία το σύστημα. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της προσπάθειας μας όλες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάπουλα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, τα καλά στατιστικά στοιχεία είναι εργαλεία αποφασιστικής ε, σημασίας για τους πολιτικούς ευθύνοντες. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε αξιόπιστα λοιπόν στατιστικά δεδομένα με μειωμένο κόστο και αντικειμενικά. Προφανώ στηρίζουμε αυτήν την ε, κατεύθυνση. Όσα μας είπαν ο εισηγητή μα και ο πρόσωπος τη Επιτροπή, νομίζω ότι καταρτίζουν μια πρόταση που ακολουθεί λοιπόν τη σωστή αυτή κατεύθυνση. Πρέπει να διασφαλίσουμε αυτήν την τάση και να υπάρχει συγκρισιμότητα στα στατιστικά στοιχεία. Διότι αν αλλάξουν οι μεθοδολογίες και είναι πολλαπλές, θα χάσουν ως προς την αξιοπιστία και την συγκρισιμότητα με τα παλιότερα στατιστικά στοιχεία. Πιστεύουμε όμως ότι από τεχνικής άποψης μπορούμε να λάβουμε τις απαραίτητες μέρημνες ώστε να οδηγηθούμε μαζί με τον εισηγητή και ε, στην σωστή, στο σωστό αποτέλεσμα. Η ομάδα μου λοιπόν στηρίζει την πρότασή του. Κύριε Μεντέλτσεβα, κάποιο σχόλιο. Ναι, ε, και για τις προηγούμενες παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ και την ομάδα των σοσιαλιστών που με στηρίζει στην όλη μου προσέγγιση. Η έκθεση φαίνεται να πηγαίνει στην ε, σωστή κατεύθυνση λοιπόν και για το πρώτο σας ερώτημα, αν υπάρχει συγκεκριμένα παραδείγματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα πλουστευτούν οι πίνακες. Ε, μας ε, δόθηκε ένα τέτοιο παράδειγμα, θα το μοιράσω και στα υπόλοιπα μέλη. Και είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου το εξή, ότι περνάμε από μια εκατοντάδα πινάκων σε μια δεκάδα πλέον. Γι' αυτό μιλάμε για πλούστευση. Και κάτι άλλο που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι η Επιτροπή ασχολήθηκε και με το θέμα των ορίων, των κατοφλίων. Μέχρι τώρα ήταν διαφορετικά τα κατόφλια. Δηλαδή, οι εκμεταλλεύσει μικρών διαστάσεων δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είχαμε και μικρή ποσότητα παραγωγή. Τώρα με τον νέο κανονισμό δεν πάμε προ ομοιογενειοποίηση, κάτι που φαίνεται να ανησυχεί τον συνάδελφο Ντόρφμαν, αλλά αυτό που στοχεύουμε είναι να έχουμε περισσότερη αντιπροσωπευτικότητα για να γνωρίζουμε καλύτερα τι περιφέρειέ μα, τι περιοχέ, τι προσδοκίε των παραγωγών και ανάλογα με τα μέτρα που λαμβάνονται να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες απλών προτάσεων. Έχω λοιπόν καταγράψει τα διάφορα επιχειρήματα που υπάρχουν από όλε τι πλευρέ. Ευχαριστώ του συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση και θα τα λάβω υπόψη όλα στο μελλοντικό σχέδιο έκθεση. Θα ευχαριστήσω επίση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι ιδιαίτερα εντελεχεί απαντήσει τη και Υπήρχε μια έκφραση που ακούστηκε εδώ, το δικαίωμα παρακολούθηση ε, εξέταση των θεμάτων τη Γεωργία από το Ευρωκοινοβούλιο. Να θυμίσω ότι με τη συνθήκη τη Λισαβόνα δεν είναι απλώ δικαίωμα ε, παρατήρηση εδώ. Και σε κάθε περίπτωση θα ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικοδομητική τη στήριξη στην προετοιμασία τη εκθέση. Ευχαριστώ και του συναδέλφου. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό. Να θυμίσουμε λοιπόν στην Επιτροπή ότι έχουμε εξουσία συναπόφασης εδώ. Υπάρχει βεβαίως ε, καθεστική ατάξη μετά από μια το, ιστορία τόσων ετών και τέτοια παράδοση, όμως το Ευρωκοινοβούλιο θα καταλάβει το χώρο που το αρμόζει πλέον. Περνάμε στο επόμενο σημείο, ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση, σχετικά με την κατάσταση των τομέων των πουλερικών και των αυγών. Πρώτα απ' όλα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Williams με μια σύντομη παρουσίαση του κύριου Στικ, Προέδρου των Ευρωπαίων Μερμπορών Αυγών, Πουλερικών και Προϊόντων σχετικών. Κύριε Στικ, έχετε το λόγο. Herr er- Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω την Επιτροπή, η οποία μα προσέφερε τη δυνατότητα να αναφερθούμε στην ε, νέα οδηγία 499 για να δώσουμε τι τις εκτιμήσεις μας για τις μέχρι τώρα εξελίξει ε, για την ισχύουσα κατάσταση και να κάνουμε προτάσει ε, για τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουμε ότι θα πρέπει στο μέλλον να εξελιχθεί η κατάσταση. Έχουμε περιορισμένο χρόνο στη θέσή μας και γι' αυτό προχωρώ δίνοντας το λόγο στο Γενικό Γραμματέα κύριο Μαρκ Βίλιαμς για να σας κάνει την παρουσίαση και τις, ε, να εκφράσει απόψεις μας. Παρακαλώ. Ο κύριος Βίλιαμς λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι. Θα ήθελα να σας δείξω εννέα διαφάνειες οι οποίες μας δείχνουν ε, επίκαιρα και αντικειμενικά στοιχεία για την κατάσταση μετά από την εφαρμογή της οδηγίας για την ευημερία των οτοκών ορνήθων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιομηχανία αυτή από το 1999 προσπαθεί να υλοποιήσει σωστά την οδηγία. Την οδηγία μάλλον ε, το 1999 και εδώ αυτό που πρέπει να να εξασφαλίσουμε όπως με κάθε νομοθεσία θα αποφύγουμε τα προβλήματα. Σε γενικές γραμμές είναι η μεγάλη παραγωγή στα περισσοτερα κάτι κράτη-μέλη, αυτοί που θα μπορέσουν να ανατηρήσουν τις προθεσμίες για την απαγόρευση των συμβατικών κλοβών μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012. Πιστεύουμε ότι οι μικρότεροι παραγωγοί δεν θα τα καταφέρουν ή θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν αυτή την, την αγορά, αυτόν τον τομέα. Ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι για να σας ενημερώσουμε, να σας πούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανησυχίες, ποια είναι, ποια είναι η αναλογία με το πέρασμα σε διεθετημένους κλοβούς ή συστήματα που δεν χρησιμοποιούν κλοβούς για την παραγωγή και τι ακριβώς συμβαίνει με την ε, συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τα αυγά που παράγονται σε συμβατικές κλοβούς, σε σημαντικούς κλοβούς δεν θα τίθενται στην αγορά από 1η Ιανουαρίου 2012. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μεγάλη έλλειψη σε αυγά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρξει και σημαντική αύξηση στην τιμή των αυγών. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρξει συστηματική μετακίνηση προ τα συστήματα τα διευθετημένα ή συστήματα που δεν χρησιμοποιούν κλοβού. Οι επόμενε τρει διαφάνειε νομίζω δείχνουν το πρόβλημα σε όλε τι διαστάσει. Όπως βλέπετε από το διάγραμμα, με πράσινο έχουμε τον αριθμό των ε, ορνήθων που βρίσκονται στα συμβατικέ κλωβούς το 2008. Το κίτρινο δείχνει τα συστήματα σε κοτέτσια, το άλλο της ελευθέρας βοσκής και έπειτα τους διευθυντημένους κλωβούς. Η ελαφρά πράσινη το ελαφρά πράσινο κομμάτι του διαγράμματο δείχνει στοιχεία από την Γενική Διεύθυνση Γεωργία από το 2008 και αποδεικνύει ότι 19 περίπου εκατομμύρια ε, όρνηθες από τα 354 του συνολικού αριθμού ορνήθων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βρίσκονται σε διαθετημένους κλωβούς. Το 1999 βλέπουμε ότι έχει μειωθεί κάπως η περιοχή των συμβατικών κλοβών. Η κίτρινη και η πράσινη περιοχή λοιπόν έχουν μειωθεί κάπως και περισσότερες ορνήθες έχουν περάσει σε διαθετημένους κλωβούς. Βλέπουμε ότι έχουν μεγαλώσει κάπως οι αναλογίες των ελευθέρας βοσκής, των βιολογικών και των εκτατικής εκτροφής ορνήθων. Τώρα περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η πρόβλεψή μας για το 2012. Βλέπουμε ότι η πράσινη περιοχή και οι πράσινοι με άσπρα στίγματα έχουν ε, μειωθεί. Αλλά αυτό που μας απασχολεί είναι η πράσινη περιοχή. Προβλέπουμε ότι εκεί θα υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια όρνηθες που δεν θα συμμορφώνονται με την νομοθεσία ε, μέχρι το 2012. Αν το υπολογίσουμε αυτό σε σχέση με το συνολικό αριθμό ορνήθων, 353 εκατομμύρια, είναι περίπου το 29% του συνολικού αριθμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν διαμορφώνονται δύο πιθανότητες έως το 2012. Δύο σενάρια. Η Επιτροπή λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν την απαγόρευση για τις συμβατικές κλωβούς. Εμείς συμφωνούμε απολύτως με αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι εάν οι αριθμοί μας είναι σωστοί, δηλαδή θα πρέπει να πετάμε 83 εκατομμύρια αυγά την ημέρα. Αν αυτό συμβεί, η ευρωπαϊκή αγορά και οι καταναλωτέ θα στηριχθούν 83 εκατομμύρια αυγά την ημέρα. Επειδή είναι πολύ αυστηρή η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Σαλμονέλα, υπάρχουν μόνο τρει χώρες εκτός Ευρώπης που έχουν την εξουσιοδότηση να πολλούν τα ολόκληρα αυγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελβετία, η Κροατία και η Νορβηγία συγκεκριμένα. Επίση, η αγορά προφανώ υπόκειται στου κανόνε τη αγορά και τη ζήτηση. Τη προσφορά και τη ζήτηση, συγγνώμη. Αν λοιπόν υπάρχει έλλειψη στην προσφορά, θα υπάρχει και αύξηση των τιμών. Και αυτό σημαίνει ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η ευρωπαϊκή παραγωγή μπορεί να αντικατασταθεί από εισαγωγέ αυγών και προϊόντων αυγών, που θα προέρχονται όμω από παραγωγού με χαμηλότερε προδιαγραφέ για την ευημερία των ζώων. Αυτό δεν πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει την ευημερία των οθόκων ορνήθων, τους καταναλωτές, την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ε, καλλιεργητές μετριακών, το περιβάλλον και την ε, επιστημιστική ασφάλεια, καθώς και την οικονομία. Η άλλη τώρα πιθανότητα, το άλλο σενάριο είναι ότι αν υπάρξει αρκετό χρόνο προκειμένου να συμμορφωθούν τα κράτη-μέλη, δηλαδή αν δεν εφαρμόσουν την νομοθεσία τα κράτη-μέλη αυστηρά, τότε θα συνεχιστεί η παραγωγή από συμβατικέ κλοβού και αυτό στην αγορά σημαίνει ότι θα υπάρξουν σοβαρέ ε, διακοπές. Δηλαδή, η βιωσιμότητα των ε, ένομων των επιχειρήσεων που παρακολουθούν τον, ε, την νομοθεσία θα, η δραστηριότητα του θα πληγεί. Αυτό σημαίνει ότι και η παραγωγή των κλωβών θα πληγούν. Και όλα τα συστήματα παραγωγής, είτε είναι σε κλωβούς, είτε εκτατικά, είτε ελευθερασβοσκής, είτε βιολογικά. Και επίση είναι άδικο για του παραγωγού που θα έχουν επενδύσει ε, στη λήψη μέτρων για να συμμορφώνονται με την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί λοιπόν πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση και ελπίζω να μου δώσετε την ευκαιρία να σα τα εξηγήσω τα τη διαφορετική προσέγγιση. Για μα είναι πολύ σημαντικό για την αγορά αυτή και για όλου όσου παράγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφύγουμε την έλλειψη αυγών ε, εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και την σημαντική αύξηση των τιμών. Ωστόσο, είναι ένα αναντήρητο γεγονό ότι αν μελετήσει κανεί του αριθμού όπω του έχουμε δει ω τώρα και αν θεωρήσουμε ότι είναι ακριβεί οι προβλέψει μα, σίγουρα κάποια Ευρωπαϊκή παραγωγή δεν θα είναι έτοιμη για την απαγόρευση των συμβατικών κλοβών. Εάν λοιπόν οι νομοθέτε και οι πολιτικοί θύνοντες αφήσουν περισσότερο περιθώριο χρόνου, τότε πιστεύουμε ότι θα χρειαστούμε ένα κύκλο ή δύο κύκλους παραγωγής αυγών από τις οτόκες όρνηθες για να προσαρμοστούμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πυκνότητα των κοπαδιών ε, των ε, ορνήθων και να λάβουμε υπόψη την ε, ανάγκη σε έκταση 750 εκατοστά ανά όρνηθα και να, δούμε τι θα γίνει και με τα επιτραπέζια προϊόντα. Διότι εάν δεν ληφθούν αυτά τα απαραίτητα μέτρα, παραγωγοί δεν θα μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα του σε άλλα κράτη-μέλη και αυτό θα πλήξει του παραγωγού του δεύτερου κράτου-μέλου, του λόγω κράτου-μέλου. Εάν οι παραγωγοί λοιπόν έχουν λίγο περισσότερο χρόνο, θα πρέπει να έχουν ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα για να ξέρουν πώ μπορούν να περάσουν σε ένα διαθετημένο σύστημα ή σε ένα σύστημα χωρί κλοβού. Αυτό θα πρέπει να το εγκρίνει αρμόδια εθνική αρχή. Και θα δώσω ω παράδειγμα την Γερμανία όπου θα απαγορευτούν οι συμβατικέ κλοπέ λίγο νωρίτερα. Εκεί πρέπει να υπάρχουν αυστηρέ κυρώσει ε, για όσου δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία. Το άλλο καθοριστικό ζήτημα είναι η επιβολή της νομοθεσίας. Όπως ε, ξέρετε, ένα αυγό είναι αυγό. Δηλαδή δεν μπορεί κανεί να πει τη διαφορά μεταξύ των συστήματων, συστήματων παραγωγή, να δει ποια είναι η διαφορά μεταξύ των συστήματων παραγωγή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει κάποιο μέθοδο για τη διάκριση των αυγών όπω παράγονται από συμβατικέ κλωβού ή από τα άλλα συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι τα μόνα αυγά που νομίμω θα μπορούν να τίθενται στην αγορά από 1η Ιανουαρίου είναι αυτά που προέρχονται από διευθετημένου κλωβού. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και ειδική μέρημνα γι' αυτό, αλλά αν δοθεί περισσότερο χρόνο στους παραγωγούς θα χρειαστεί μια διαφορετική ένδειξη για τα αυγά που θα συνεχίσουν να βρεχόνται από συμβατικέ κλωβούς. Ε, Ένα αριθμό, όπω ε, για τα διαθετημένα θα έχουμε τον αριθμό 3, για τα συμβατικά να έχουμε το 4 ή κάτι ανάλογο. Επίσης θα πρέπει οι ελεγκτές να αυξήσουν τις επισκέψεις επιθεώρησης για να βεβαιωθούν ως προς την υλοποίηση της νομοθεσίας. Θα πρέπει οι αρμόδιες εθνικές αρχές να αναλάβουν αυτή την ευθύνη βεβαίω και δεδομένη της διορίας που δίδεται, οι επισκέψεις αυτές μπορεί να, γίνουν, να έχουν γίνει και δύο-τρία χρόνια πριν από την πραγματική επιβολή των μέτρων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, συμπερασματικά Πιστεύουμε ότι το να μην κάνουμε τίποτα και να παραμείνουμε αδρανεί δεν είναι πλέον κάτι που μπορεί να συμβεί. Η βιομηχανία τη παραγωγή αυγών είχε 12 χρόνια στη διάθεσή τη για να εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία. Συμφωνώ ότι σε άλλε περιπτώσει θα ήταν απλό ίσω αυτό και θα μπορούσαμε να είχαμε την απέτηση να έχουν συμμορφωθεί όλοι. Όμω το 2005 η Επιτροπή και οι Υπουργοί αποφάσισαν ότι η έκθεση αυτή που καθορίζει τα συγκεκριμένα μέτρα καθυστέρησε τρία χρόνια. Αποφασίστηκε η προηγούμενη οδηγία να ισχύσει, να υπάρξει δηλαδή παράταση και βρεθήκαμε στην εξή κατάσταση. Η παραγωγή δεν θέλουν να επενδύσουν στους διεθνούς κλωβούς ε, πριν γίνει υποχρεωτική νομοθεσία. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι πιέζονται και τελευταία στιγμή αλλάζουν τους κλωβούς. Έτσι λοιπόν προσκαλούμε την Επιτροπή και εσάς να παρέμβετε, διότι αν δεν συμβεί αυτό δεν θα έχουν απομακρυνθεί εγκαίρω όλε οι όρνητε από του κλοβού. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε τι υψηλέ μα προδιαγραφέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να μην έχουμε και την εξαγωγή τη δική μα παραγωγή σε τρίτε χώρε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας το θυμίζω και συγχωρήστε με που σας το λέω. Ε, είναι γεγονός ότι πέραν της Ελβετίας όλες οι χώρες που είναι βασικοί εμπορικοί μας εταίροι για τα αυγά και τα προϊόντα αυγών δεν έχουν νομοθεσία ευημερία των ορνήθων ε, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα στα κοπάδια ορνήθων. Δεν ε, εξετάζουν καν όπως εμείς τους κλωβούς. Ε, ζητήσαμε λοιπόν από την Επιτροπή να μας πει αν είναι δυνατόν τα κράτη-μέλη να παράσχουν ε, επιμέρους δεδομένα για το τι γίνεται με τα διάφορα συστήματα παραγωγής και την ευημερία των ορνήθων, ώστε να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει στην πράξη. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Έχω και άλλε διαφάνειε να σα δείξω αν σα ενδιαφέρουν τα στοιχεία αυτά, αλλά θα σα τα διαθέσω και offline, εάν θέλετε περισσότερε πληροφορίε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Williams για την παρέμβασή του. Αρκετοί συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. Αλλά μια και γίνεται απευθεία, απευθύνθηκε μάλλον απευθεία ο λόγο και έγινε αναφορά προσωπικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρότεινα να επιτρέψουμε στον κύριο Καβινέλη πρώτα να απαντήσει, να δώσει τη σχετική ενημέρωση και στη συνέχεια όποιος επίσης θέλει να λάβει το λόγο, να έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί στο σύνολο των παρεμβάσεων, να μιλάει το κοινοβούλιο τελευταίο αυτή τη φορά. Κύριε Καβινέλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας για τη συζήτηση αυτή. Καταρχάς να διευκρινίσω ότι η Επιτροπή απάντησε σε πολλές περιπτώσεις τα αιτήματα που έθεσε όχι μόνο ο κλάδος αλλά και τα κράτη-μέλη. Τα αιτήματα αυτά διευκρινίστηκαν όχι μόνο στις διάφορες διαχειριστικές επιτροπές αλλά και στην μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή. Κάθε μήνα αναθεωρούνται τα στοιχεία τα δε αιτήματα που υπέβαλε και ερωτήματα που παρουσίασε ο κύριος Βουίλιαμς έχουν αντιμετωπιστεί και αυτά. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και για την μελέτη που διεξήγαγε για τον κλάδο της ε, αγοράς και για το μέλλον όχι μόνο για τα αυγά αλλά και για το κρέας. Μιλώ για την επιτροπή που είχε υποβληθεί στην επιτροπή αυτή τον Αύγουστο. Στα λίγα λεφτά που έχω στη διάθεσή μου θα ήθελα να αναφερθώ στην άποψη της Επιτροπής για τις συστάσεις που βρίσκονται σαν συμπέρασμα της μελέτης. Πρώτον, οι συστάσεις μιλούν για την ανάγκη να βελτιωθεί η εφαρμογή της οδηγίας. Όπως γνωρίζετε η εφαρμογή της οδηγίας αποτελεί βασική ευθύνη των κρατών μελών που έχουν την πλήρη ευθύνη της ενσωμάτωσης και εφαρμογής της. Τα κράτη-μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή τα στοιχεία των επιθεωρήσεων και ελέγχων που διεξάγουν και τα στοιχεία, τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αιτήσια κλίμακα και η Επιτροπή σπέβδει να τα αναλύσει σε μόνιμη βάση. Επιπλέον, η αρμόδια κτηνιατρική επιτροπή της, επιτροπή, κτηνιατρική επιτροπή της Κομισιόν επισκέφθηκε τα τελευταία χρόνια 20 κρατημέλη και στο μέλλον, το 2011, θα επισκεφθεί άλλα 6. Όλα αυτά βάσει και των πόρων που έχει η Κομισιόν στον τομέα της ε, ε, ευημερία των ζώων που είναι πόροι που όπως ξέρετε είναι περιορισμένοι σε σχέση με τα αυξανόμενα αιτήματα της κοινωνίας. Υπογραμμίζουμε, στο να, υπογραμμίζει λοιπόν ότι ε, οι δυνατότητες επιτροπής είναι αρκετά περιορισμένες στον τομέα αυτό. Πρόκειται για μια πολιτική επιλογή. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να αναλύσουμε και να, και να αξιολογήσουμε τι θα κάνει η Επιτροπή στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προετοιμάζει μια στρατηγική για την προστασία των ζώων που θα υιοθετηθεί το 2011 και που βασίζεται σε μια αξιολόγηση της τελευταίας 20 ετίας στην, την πολιτική προστασία των ζώων στην Ένωση. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για τις συστάσεις. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο που είχε η γρήπη των πουλερικών στην αγορά και την ανάγκη διασφάλισης ε, καθησυχασμού των ε, καταναλωτών, πρόκειται για μία από τις σημαντικές συστάσεις της έκθεσης, η Επιτροπή, όπως ξέρετε στο παρελθόν, ξεκίνησε με οικονομική υποστήριξη της δραστηριότητα αυτή, με ε, μια πολιτική διαφάνεια και μάρκετινγκ του ευρωπαϊκού προϊόντος. Κατά βάση είμαστε πεπισμένοι ότι είναι σημαντικό να εκπαιδευτεί ο καταναλωτής ε, και χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο. Την 1η Οκτωβρίου θα κάνουμε μια διάσκεψη για την ευημερία των ζώων στο Σαρλεμάνι με πάνω από 520 άτομα που θα μετέχουν. Είναι η πρώτη τέτοια διεθνή εκδήλωση. Θα μιλήσει το Κοινοβούλιο στο ξεκίνημα. Έχει δεχθεί η κυρία Πόλσεν ε, την ε, πρόσκληση να μιλήσει στην ενακτήρια συνάντηση όπως ο κύριο Ντάλι. Πιστεύουμε λοιπόν ότι και η επικοινωνία και η εκπαίδευση είναι σημαντικές. Για την σύσταση τώρα σε ό,τι αφορά την προστασία από αυγά εισαγωγής χαμηλότερης τιμής. Όπως ξέρετε, ο κύκλος διαπραγματεύσεων για τις Ντόχας ε, συνεχίζεται. Περνάει μια σημαντική φάση όπου συζητούνται όλα τα non-trade θέματα, περιβάλλον, προστασία των ζώων κλπ. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα της ευημερία των ζώων, η Επιτροπή σε όλες τις ε, διμερείς σχέσεις που έχει με οποιοδήποτε τέρο, η Κομισιόν επιμένει να, βάλει, να μπαίνει ως προτεραιότητα η ευημερία των ε, ζώων και ως ε, απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε υπογραφή ε, κτηνιατρική συμφωνία. Έχουμε πετύχει αποτελέσματα, θα συνεχίσουμε προς, τα, προς την ίδια κατεύθυνση, άρα την σύσταση αυτή τη δεχόμαστε απόλυτα και την προωθούμε ήδη. Υπάρχουν δύο ακόμα συστάσεις στο τέλος της έκθεσης. Πρώτον, σταθερή νομοθετική βάση, να μην αλλάξει δηλαδή εκ νέου η οδηγία με απόλυτη απο, ε, απαγόρευση των κλοβών στο μέλλον. Ξέρετε ότι αυτό που θα γίνει το 12 δεν είναι απαγόρευση, αλλά μετατροπή των κλοβών από παραδοσιακές σε εμπλουτισμένες. Είναι σαφές ότι μακροπρόθεσμα δεν θα χρειαστεί να αλλάξει η υφιστάμενη οδηγία. Οποιοδήποτε μελλοντικό μέλλον ε, χρειαστεί να ληφθεί θα γίνει μετά από ανάλυση του οικονομικού και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Αυτό είναι σαφές. Τελευταία σύσταση. Οικονομική υποστήριξη των παραγωγών της Ένωσης με βάση τα προγράμματα της ανάπτυξης της ε, ε, Εγώ ανήκω στη Γενική Διεύθυνση Καταναλωτών. Ασχολούμαι με την ευημερία των ζώων. Ξέρω ωστόσο τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα ε, στα πλαίσια τη ανάπτυξη ε, ανάπτυξης για την ευημερία των ζώων. Επιβεβαιώνω ότι πολύ λίγε είναι. Ελάχιστε χώρε μέλη μέχρι τώρα έχουν ζητήσει να χρησιμοποιήσουν τα μέτρα αυτά για την ευημερία των ζώων. Δαπανίσαμε πολύ λίγο σε σχέση με, την, ε, ζήτη, με το αίτημα των καταναλωτών. Η Επιτροπή λοιπόν θα συνεχίζει να απαιτεί να υπάρξει και να πιέζει να υπάρξει επίγνωση από πλευράς των, των οργάνων στα κράτη-μέλη για την ύπαρξη των μέτρων αυτών και όχι μόνο προς τα κράτη-μέλη αλλά και προς τα ενδιαφερόμενα μέρη για να υπάρξει μία προσέγγιση των, των ετοιμάτων με την οικονομική υποστήριξη. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο σε κάποιε χώρε και το δείχνει η μελέτη. Αυτέ είναι απόψεις της επιτροπή για τι πέντε συστάσεις ε, της μελέτης. Όπως είπα, η δήλωση και στη, ξέρει την δήλωση και την έρευνα του κύριου σε Επιτροπή και εμεί άλλωστε κάθε μήνα χάρη στην διαδικασία παρακολούθησης που κάνουμε μέσω του κλάδου των αγορών δίπλα μου είναι η υπεύθυνη Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καβινέλη. Θα περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις σε σχέση με τα όσα ακούσαμε. Η ώρα είναι ήδη 12. Έχουμε 12 εν όλο παρεμβάσεις στον κατάλογο. Παρακαλώ τους συναδέλφους να περιοριστούν στα δύο λεπτά παρέμβασης ο καθένας. Ξέρετε ότι πρέπει στις 12.30 να σταματήσουμε για να επιτρέψουμε τους διερμηνείς να ξεκουραστούν. Ο κύριος Κανόψικη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς τον επότροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εκ των οποίων η πρώτη έχει να κάνει με το κόστος της παραγωγής και το κόστος των ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται στην εκτροφή όρνηθας. Εισήχθη πριν από καμιά δεκαετία περίπου χρόνια η απαγόρευση της χρήσης κτηνοτροφών από οστεάλευρα ή κρέατα άλευρα. Όμως βλέπουμε εντωμεταξύ ότι από την επιστημονική έρευνα φαίνεται πως δεν έχει αποδειχθεί η ή μάλλον δεν προξενεί η χρήση κρεαταλεύρων και οστεαλεύρων ε, προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία. Ερωτώ λοιπόν τι κάνει στο θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Όταν έχουμε εισαγωγές από κρέατων από τρίτες χώρες τα οποία κρέατα έχουν εκτραφεί με ε, ζωάλευρα, κρεατάλευρα ή ε, οστεάλευρα, γιατί να υπάρχει απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της χρήσης τους. Και επίσης γνωρίζουμε ε, ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν εισαγάγει νέα τεχνολογία που επιτρέπει τον περιορισμό των οτόκων ορνήθων και της παραγωγής. Ωστόσο, με δεδομένη την εξέλιξη στην ε, ε, ζήτηση και την αγορά μπορούμε να περιμένουμε μια ικανοποιητική κατάσταση για τα επόμενα χρόνια στον χώρο της ορθινοτροφίας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σαφέστατη ερώτηση. Ο κύριος Λάιονς και παρακαλώ σύντομα για τον έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. θέλω να πω ότι δεν μπορούσα να φανταστώ τόση πια ικανοποίηση, αυταρέσκεια, ευχαρίστηση από όλα αυτά που μας παρουσιάζεται σε ένα θέμα τόσο σοβαρό, σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί και προβληματίζει τόσους παραγωγούς στην Ευρώπη που έχουν επενδύσει εκατομμύρια στην παραγωγή. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πώς οι επενδύσεις τους δεν θα υπονομευθούν Το μικρόφωνο του μιλτή δυστυχώ δεν είναι αναμένο σωστά, δεν ακούγεται καθαρά. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μία προσπάθεια. Να έχουμε λοιπόν ένα ποσοστό αναμετατροπής αρκετά σημαντικό, το οποίο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί εν μία νυχτή. Μέσα στους επόμενους μήνες λοιπόν δεν πρόκειται να λυθεί το ζήτημα αυτό και παρακαλώ την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα θέματα σοβαρά και να εισακούσει τις παρατηρήσεις των Ευρωπαίων παραγωγών. Ευχαριστώ, Τζορτζ. Σε φέστατα τόσο είπες. Είναι πραγματικά σημαντικό το θέμα αυτό για μα. Γι' αυτό το, προβλά... το προβλέψαμε στην ημερήσια διάταξη και μα ευαισθητοποιεί ιδιαίτερα. Γι' αυτό και αναζητήσαμε μια απόκριση και θέλουμε μια απόκριση που να μην είναι γενικόλογη. Το πρόγραμμα υπάρχει. Υπάρχει γιατί ακούσαμε και του εκπροσώπου του τομέα αυτού και ένα μεγάλο μέρο των παραγωγών δεν είναι έτοιμο να συμμορφωθεί με την νομοθεσία. Δεν μπορεί να αναβάλλεται όμω συνεχώ η επίλυση του προβλήματο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει εν γέννη συμφωνία σε επίπεδο επιτροπής μας ε, για όλο το θέμα αυτό. Από την προηγούμενη συνεδρίαση που ήταν κάπως ε, πιο δυσάρεστη. Θα προσπαθήσω εγώ τώρα να είμαι κάπω πιο συμφιλιωτικός, ελπίζοντα ότι θα μπορέσουμε όμως να βρούμε λύσεις ικανοποιητικές και για τους παραγωγούς. Ε, με εντυπωσιάζει και με παραξενεύει η πρόταση της Επιτροπής, γιατί νόμιζα ότι είχαμε συνεννοηθεί μεταξύ μα ότι θέλουμε να ε, προαγάγουμε υψηλέ προδιαγραφέ εκτινοτροφία. και ότι έχουμε συμφωνήσει σε αυτές. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει και τέτοια μέσα στη διάθεσή της, δεν, είναι, δεν έχει τη, τη διάθεση να τα αξιοποιήσει. Μας είχατε διαβεβαιώσει ότι θα, εισάγα, θα εισάγατε μια ε, διακοινωτική απαγόρευση και ότι θα φροντίζατε να τιμωρηθούν τα κράτη τα οποία δεν ε, ακολουθούν αυτή την απαγόρευση. Και τώρα βλέπω ότι αρνείστε να τηρήσετε αυτά που έχετε υποσχεθεί. Μπορείτε να μα πείτε ποια είναι τα κράτη στο Συμβούλιο τα οποία δεν συνεργάζονται. Επίση, όταν μα λέτε ότι 80 εκατομμύρια αυγών ξαφνικά γίνονται παράνομα, τι είναι αυτό. Τι σημαίνει αυτό, μια μεγάλη διάσκεψη για την ευημερία των ζώων στο Σαρλεμάνια τις προηγούμενες μέρες που έγινε. Δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα. Γι' αυτό παρακαλώ λοιπόν να είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι και πιο, ε, να έχουμε πνεύμα συνεργασία στην υπόθεση αυτή. Αλλά επαναλαμβάνω δεν καταλαβαίνω γιατί η Επιτροπή δεν θέλει να ε, ανταποκριθεί στα όσα έχει, στις δεσμεύσεις τις οποίες έχει ήδη αναλάβει. 83 εκατομμύρια αυγά την ημέρα δεν, μπορούμε, δεν μπορούν να καταστραφούν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε μία λύση. Τα αυγά τα οποία δεν θα πληρούν τις προδιαγραφές που ουσιαστικά θα είναι παράνομα και θα αναγνωρίζονται, θα ταυτοποιούνται ω τέτοια, θα πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε και οι παραγωγοί που τα έχουν να μην βρίσκονται σε δύσκολη θέση, να μην τιμωρούνται χωρί λόγο. Πρέπει να βρούμε μια λύση, μια ερμηνεία διαφορετική τη νομοθεσία. Και αν η νομοθεσία δεν είναι καλή και πρέπει να τροποποιηθεί, ε, αυτό θα κάνουμε ω κοινοβούλιο δημοκρατικά ελεγμένο. Εμεί ε, που είμαστε εκλεγμένοι από του ψηφοφόρου, εσεί που θέλετε να επιβάλλετε κάποιε συγκεκριμένε προδιαγραφέ, στι οποίε είμαστε και εμεί σύμφωνοι, θα συνεργαστούμε για να κάνουμε μια τροπολογία, μια τροποποίηση νομοθεσία. Αλλά πείτε μα ποιε είναι οι προδιαγραφέ, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν αυξήθηκαν οι απαιτήσει από τους παραγωγούς της Ένωση δεν ξέραμε για την ύπαρξη της κρίσης, της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της κρίσης που αντιμετώπιζε με τόσο δραματικό τρόπο η Ευρώπη, ούτε και ξέραμε πώς θα επηρεάσει την παραγωγή η τιμή των σιτηρών. Καταλαβαίνω ότι πολλοί είναι οι λόγοι που οδηγούν στην καθυστέρηση της διαδικασίας αλλαγής των νέων κλοβών και ότι οι νέες δομές δεν έχουν γίνει, οι νέες, τα νέα πλαίσια δεν έχουν γίνει ε, σωστά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το ότι εισάγουμε αυγά από κλοβούς που είναι χειρότερη κατάσταση από τους δικούς μας και βοηθάμε παραγωγούς ξένων χωρών για να το κάνουν αυτό. Μα δεν καλύτερα να το κάνουμε βοηθώντας τους ε, Ευρωπαίους παραγωγούς. Αν είμαστε και λίγο ευέλικτοι θα καταλάγαμε, θα καταλαβαίνουμε ότι και οι αντίστοιχε χώρες ε, είναι εξίσου ευέλικτοι ε, από όσο και οι δικοί μας. Συνεχίζουμε να εισάγουμε προϊόντα από ε, ε, κλοβούς χειρότερης ποιότητας. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε όμως για ένα τόσο σημαντικό θέμα μόλις δύο λεπτά. Είναι δυνατόν για ένα θέμα για το οποίο η Επιτροπή μπόρεσε ε, να φλιαρίσει επί 15 λεπτά χωρί να μα πει ουσιαστικά τίποτα. Έχω να επισημάνω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα ζήτημα αξιοπιστία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εκδίδουμε νομοθεσία, αφήνουμε περιθώριο 10 χρόνια για την εφαρμογή τη και τώρα έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια τελείω χαλαρή προσέγγιση και τιμωρεί ουσιαστικά εκείνου οι οποίοι έχουν επενδύσει στην εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία και δίνει πλεονέκτημα σε εκείνου οι οποίοι περίμεναν απλώ χωρί να πράξουν τίποτα, έμειναν να δρανίσουν αυτά τα χρόνια. Έχω ρωτήσει από την προηγούμενη φορά τρει συγκεκριμένε ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη ήταν τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Απλώς θα χαρακτηριστούν παράνομο όλα αυτά, θα έχουμε δηλαδή μία ε, δίκη μία προσφυγή στα δικαστήρια η οποία θα κρατήσει χρόνια και θα τραβήξει επιμακρών χωρί να βρίσκει κανεί τη λύση ή θα προχωρήσουμε σε μια διαφορετική ερμηνεία ή εφαρμογή τη νομοθεσία. Δεύτερον, πώ μπορούμε να ενημερώσουμε τον καταναλωτή για τι υψηλέ προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χαμηλότερε προδιαγραφέ που ισχύουν στην παγκόσμια αγορά. Και τρίτον, και πάλι δεν έχω λάβει στην, στην ερώτηση αυτή απάντηση, πώς μπορούμε τη νέα κοινή γεωργική πολιτική να την αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να στηρίξουμε εκείνου του παραγωγούς οι οποίοι το όντι τηρούν τις προδιαγραφές και την αυστηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ερωτώ λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί, θα ε, πήγαινα να πω να βραχεί εν πάση περιπτώσει, να βάλει το πόδι στο νερό. Αλλά δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή την, ερώτηση, την, έκφραση. Εν πάση περιπτώσει νομίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί να αποτολμήσει την αποκοτιά, να έρχεται και να ανατρέπει αυτά τα οποία μα έχει πει. μα. έχει ενημερώσει ήδη μία φορά και τώρα επανέρχεται. Μα γελιοποιεί ουσιαστικά χωρί να απαντά καν σε ερωτήσεις μας. Και εγώ θα έλεγα το εξή είναι πολύ απλό. Μαζί με του αδέρφου από την Επιτροπή του περιβάλλοντο, να καταθέσουμε μια κοινοβουλευτική επερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίπεδο ολομέλεια. πράγμα το οποίο απευθύνεται πλέον στον Επίτροπο και έτσι ο Επίτροπος είναι υποχρεωμένος να έρθει στην Ολομέλεια και να μας να δείξει και ενώπιον, μπροστά, ε, ενώπιον όλου του κόσμου και να δείξει ότι δεν, ε, ε, είναι, δεν βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι στα ζητήματα των ζωοτροφών χρειάζεται πλέον να ορθώσουμε το ανάστημά μας. Πριν από δύο χρόνια ακόμη ως συντάκτης ε, της έκθεσης από την Επιτροπή του Προϋπολογισμού των Προϋπολογισμών είχα πει ότι χρειάζεται η επαρκής υποστήριξη της αποκεντρωμένης υπηρεσίας ζωοτροφών ε, και τροφών. Ε, το Συμβούλιο ξέρουμε ότι είναι αντίθετο στι προτάσει μα και το δεχόμαστε έστω. Ξέρουμε με ποιον έχουμε, να αντιμετωπίσουμε. Αλλά η Επιτροπή υποτίθεται ότι είναι με το πλευρό μα. Δεν θα έπρεπε να κάνει κάτι περισσότερο. Με τη στάση που τηρεί, εγώ πραγματικά αμφισβητώ τι ίδιε τι προθέσει τη. Και παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να αλλάξει τη στάση τη, γιατί δεν θα δεχθούμε να μα γελιοποιεί κανεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντελάνου. Συμμεριζόμαστε τι απόψει. Η κυρία Μαγκίνε και μετά ο κύριο Ντότ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ φαίνεται να περπατάμε πάνω σε αυγά σχεδόν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση και με την ανοχή των συναδέλφων νομίζω δεν έχουμε Ελλάδα από την Επιτροπή τις απαντήσεις που μας αξίζουν. Η ποιότητα της παρουσίας που μας έγινε από τους Ευρωπαίους παραγωγούς αυγών μας οδηγεί στην απέτηση να θέλουμε τις απαντήσεις που μας αξίζουν. Θέλουμε προτάσεις και λύσεις. Και πολλές φορές συνομιλήσαμε τηλεφωνικά συνάδελφοι. Το ξέρετε, θα υπάρχουν ένα εκατομμύριο, εκατομμύρια παράνομες ε, κότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη να θα αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Μπορεί να υπάρξει έλλειψη στην αγορά αυγών, όμω η βασική ανησυχία είναι η εξή. Πώ εμεί ω βουλευτέ θα δεχτούμε να καταστρέφονται 83 εκατομμύρια αυγά από 1η Ιανουαρίου 2012 την ημέρα. Εδώ λοιπόν για σκοπούς προδιαγραφών ευημερία ξέρουμε ότι κάποιοι παραγωγοί ήδη έχουν κάνει τι απαιτούμενε επενδύσει, κάποιοι όχι για διαφορετικού λόγου, αλλά εμεί ω νομοθέτε μαζί με την Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσουμε με το πρόβλημα που σα ανακύπτει. Δεν έχουμε λάβει απαντήσει στι προτάσει που κάναμε και πρέπει να τις λάβουμε οπωσδήποτε. Η βασική μου μέρημνα, και νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ότι ενώ μιλά για σύγκληση εγκαταστάσεων και συμμόρφωση με του κανόνε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεχνάει ότι κάποιοι παραγωγοί πρέπει να χτίσουν νέε εγκαταστάσει, να διαμορφώσουν τι υποδομέ. Η σύγκληση λοιπόν ε, γίνεται την ίδια ώρα με τον εγγενιασμό των συστημάτων διαθετημένων κλωβών. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα από αυτό στην αγορά. Υπάρχει κατάρρευση τη αγορά αυγών σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό δεν μα έχει απασχολήσει ακόμη ω ζήτημα. Θα συμφωνήσω λοιπόν με την άποψή σα ότι αυτό το πραγματικό πρόβλημα για του παραγωγού και για του καταναλωτέ θα πρέπει να εξεταστεί σε υψηλότερο επίπεδο, στην Ολομέλεια. Εκτός και αν λάβουμε άμεσες και ε, ε, ευθυ... ευκρινείς απαντήσεις στις απαντήσεις που θέσαμε. Και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε. Κύριε Μακίνε και κυρία Ντότ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω απλώ ότι συμμερίζομαι τις απόψει μάλλον τις... Ε, τα συναισθήματα και τις απόψεις των συναδέλφων όπως τα εξέφρασαν και να πω ότι η Επιτροπή φαίνεται συνεχώς να μας απομονώνει από το ζήτημα αυτό και από την εξέτασή του για μας ως ε, βουλευτές <clears throat> σημασία έχετε εκπροσωπούμε πραγματικούς ανθρώπους, πραγματικούς παραγωγούς που είναι ε, παρόντε στι εκλογικέ μα περιφέρειε. που να γυρίσουμε στι χώρε μα και να του μιλήσουμε, να του εξηγήσουμε τι συμβαίνει. Για την ώρα τι να του πούμε, ότι η Επιτροπή κρύβει το κεφάλι τη στην άμμο Αστροφοκάμιλος και παπαριστάνει το πρόβλημα δεν υπάρχει. Δεν μα δίνει δηλαδή καμία απάντηση. Στην προηγούμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή είχα θέσει μια σειρά ερωτημάτων, όπως και άλλοι συνάδελφοι, και δεν έλαβα καμία απάντηση. Ούτε σε αυτά τα ερωτήματα. Θα ρωτήσω ξανά λοιπόν σήμερα και πραγματικά θα το εκτιμούσα αν μπορούσατε να μας δώσετε μια πραγματική απάντηση σε κάποιο από αυτά τα ερωτήματα. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 1η Ιανουαρίου 2012, όταν θα βρεθούμε στην δυσάρεστη αυτή θέση, τόσα πολλά αυγά που παράγονται στην Ένωση να παράγονται παρανόμως. Θα περάσουμε σε ένα σύστημα ελε... απαγόρευσης και πολλαπλών ελέγχων και μετά από μια τριετία θα αναλυθεί πραγματική δράση, διότι τότε η παραγωγή που εγώ λόγω χάρη εκπροσωπώ, παραγωγού του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν κάνει τις αλλαγέ που απαιτούνται, θα τους ε, θέσει σε θέση μειονεκτική ε, ως προς τον ανταγωνισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να μα λέει ότι δεν κοιτάμε το θέμα του θέμα του ΙΑΘΕ τον ανταγωνισμό και κοιτάμε μόνο την ευημερία των ζώων, αφόσον μιλάμε για υψηλέ προδιαγραφέ ευημερία των ζώων. Άρα ότι οι παραγωγοί πρέπει να επενδύουν σε συγκεκριμένε εγκαταστάσει, τότε έχουν μειονέκτηση σε σχέση με αυτού που δεν έχουν επενδύσει. Λόγω κόστου. Θα πρέπει λοιπόν να μα απασχολήσει την δικαιωτική απαγόρευση για την ε, εμπορία τέτοιων αυγών τι εγγύησει μπορεί να μα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το όλο αυτό θέμα δεν θα μεταβληθεί κι άλλο στην όλη διαδικασία. Οι διευθετημένοι κλοβοί απαιτούν τεράστιες επενδύσεις από τους ανθρώπους στην πράξη. Πρέπει να έχουν και αποζημίωση, απόσβεση των εξόδων τους και χρόνο για να τα καταφέρουν να προσαρμοστούν. Και ποιος ξέρει αν στο μέλλον δεν τους ζητηθεί να κάνουν, κι και άλλες αλλαγές. Πρόεδρο, είναι πολύ σημαντικό να προλάβουμε να δώσουμε το λόγο και πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό, επειδή έχουμε και άλλου αγροτέ, σα παρακαλώ να είσαστε πάρα πολύ σύντομοι. Η κατάσταση είναι ήδη σαφή. Πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι καιρός που περιμένουμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ ως ε, παραγωγός αυγών θέλω να δηλώσω το ιδιαίτερο συμφέρον που έχω για το θέμα αυτό. Έχουμε μια πρόταση λοιπόν, την οποία δεν ξέρω αν θα την υποστηρίξουν όλοι. Έχουμε μια σειρά από προβλημάτων που αναζητούν λύση χρόνια τώρα και για λόγους προτιμήσεως ε, των καταναλωτών τα, η παραγωγή φεύγει πλέον από τους μαζικούς κλουβούς και προχωρεί σε άλλα συστήματα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να παρεμβάσει προσδιορίζοντας στη συνέχεια μια 100% ε, μετατροπή μέσα σε πολύ στενές προθεσμίες. Πολύ καλά, έγινε όμως μια προσπάθεια να αλλάξουν τα πράγματα μέσα σε συνθήκες πολύ στενές. Όταν η βιομηχανία θεωρούσε ότι, ο κλάδος μάλλον θεωρούσε ότι, μια, ότι θα ιτηρηθούν ε, ότι δεν πρόκειται να τηρηθούν ε, οι ε, νομοθετικές διατάξεις ε, και θα μπορούσε να βρει μία διέξοδο χάρη στην πίεση των λόμπι. Ταυτόχρονα όμως έχουμε δαπανίσει το ευρωπαϊκό στο Ηνωμένο Βασίλειο 500 εκατομμύρια ευρώ του δικού μας προϋπολογισμού για την αναμετατροπή. Η τεχνητή αυτή προθεσμία οδηγεί τελικά σε δυσμενέστερες συνθήκες για εκείνους οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί στη νέα νομοθεσία και ευνοεί μόνο εκείνους οι οποίοι την αγνόησαν. Χρειάζεται να αναγνωριστεί ότι έχουν χορηγηθεί ακόμη και αναπαραγωγό μέχρι και 600.000 ευρώ ως επιδότηση χωρίς να υπάρχει συνθήκη της χρηματοδότησης. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει μέσα σε συνθήκες κρίσεως και διεπιστηστικής να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναγνωρίσει καταρχάς ότι υπάρχει πρόβλημα, ευτυχώς με υποστηρίζουν και άλλοι συνάδελφοι αυτήν την ιδέα. Δεύτερον θα πρέπει οι διατάξεις να είναι, υποστερο... να είναι ε, υποχρεωτικές και να υπάρχουν σαφείς διατάξεις για το τι, τι σημαίνει κλωβός. Δεν μπορούμε επίσης να επιτρέπουμε την ε, μεταφορά των ε, ε, αυγών αυτών από τη μία χώρα στην άλλη με τόσο, μεγάλο κόστος, τόσο διαφορετικό μάλλον κόστος παραγωγής και επίσης Υπενθυμίζω ότι η Βρετανία είναι καθαρό συνεισφορέα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και έχει δώσει χρήματα για να βοηθήσει αυτέ τι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμετατρέψουν την παραγωγή αυγών του και δεν μπορεί να επιτρέψει αυτά τα αυγά τα πιο φτηνά από τι άλλε χώρε να έρχονται στην Βρετανική αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Ο κύριος Νίκολσον. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Πάρα πολύ σύντομο θα είμαι, γιατί θέλω να ακούσω και εγώ την Κομισιόν, κυρίως αυτά που θα μας πει. Θα τους δώσω ωστόσο την ευκαιρία να μην μας πούν τίποτα. Είμαι 20 χρόνια εδώ και πρόκειται για την χειρότερη παρουσίαση που έχω ακούσει και έχω ακούσει και πολλές κακέ, αλλά πραγματικά ήταν η χειρότερη. Και πρέπει να σας πω, αν ήταν υπάλληλό μου θα τον είχα διώξει χρόνια στον εκπρόσωπο της Επιτροπής τα λέω αυτά. Νομίζουν ότι μπορούν να μας έρχονται και να μας αντιμετωπίζουν έτσι όπως μας αντιμετώπισε ο Κύριος αυτός. Εάν δεχτούμε κάτι τέτοιο πρόεδρε, το αξίζουμε. Δεν θα θέσει ερωτήσει. Τέθηκαν πολλές. Σας κάνω όμως μία πρόταση, Πρόεδρε. Να πάρετε το, το θέμα αυτό στην επόμενη συνάντηση των ιστών, να το συζητήσετε και με τους συναδέλφους στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, προχωρώντας το ζήτημα αυτό. Δεν πρέπει να τελειώσει το θέμα εδώ. Δεν μπορεί να έρχεται ε, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής και να γυρίσει πίσω και να λέει «Κοίτα, πάλι τους κατάφερα» πρόκειται για ένα θέμα πολύ σοβαρό για πάρα πολλούς. Πρέπει να τύχει καλύτερης αντιμετώπισης. Ευχαριστώ. Σίγουρα, σίγουρα. Η κυρία Πόλσον και μετά βλέπω. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. Δέκα χρόνια πέρασαν από την προηγούμενη απόφαση. Δεν μπορούμε να υπονομεύσουμε την κατάσταση λέμε, λέγοντας ότι η νομοθεσία δεν ισχύει πλέον. Θυμηθείτε ότι πάνω από το 70% της παραγωγής αυγών της Ένωσης δέχτηκαν την ανάληψη δαπανών για τις επενδύσεις που τους απαιτήσαμε. Δεν μπορούμε να τους φτύσουμε. Μια πρακτική λύση θα ήταν να πούμε ότι απαγορεύεται να παίρνουμε αυγά από τους συμβατικούς, να, να πολλούνται αυγά από τους συμβατικούς κλοβούς έξω από τη συγκεκριμένη περιοχή. Που, αλλά άλλο είναι να υπάρχει τελείως διαφορετική γραφειοκρατική αντιμετώπιση. Ο κύριος Μάγερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολλά τα θέματα. Κάποια είναι πολύ σημαντικά τα οποία, και για τα οποία θέλουμε οπωσδήποτε απάντηση από την Επιτροπή. Πρώτον, μέσα σε ένα τρίμηνο ή το πολύ ένα χρόνο θα έχουμε αυγά από κλωβούς που δεν θα επιτρέπεται να καταναλωθούν. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα γίνει η επισήμανση αυτών των αυγών ως παράνομων. Χρειάζεται για τον παραγωγό μια διαφορετική ταξινόμηση. Ας μην κάνουμε διακρίσεις με κόκκινες φραγίδες και δεν ξέρω τι, αλλά ας έχουμε κάποια σαφή ε, έτη και τοθεσία για τον καταναλωτή. Αυτό το οποίο πιστεύω δεν πρόκειται να ε, είναι και ιδιαίτερα επιβαρυντικό ή να σημάνει πολύ, πολλά έξοδα ή γραφειοκρατία, αλλά πάντως θα είναι σαφής ε, ένδειξη, θα υπάρχει μια σαφής ένδειξη. Επίσης, Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή της κατάστασης, όχι όμως με μια απλή δήλωση από τα κράτη-μέλη, η οποία δεν, έχει καμία, δεν βλέπει καμία συνέχεια για το να δίνουν τα κράτη-μέλη μια ενημέρωση που μπαίνει σε κάποιες στατιστικές και χωρίς ε, περαιτέρω ε, παρακολούθηση ή έλεγχο, απλώ μα γελιοποιεί. Άλλη παρατήρηση λοιπόν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ερώτηση: Πώ θα επαληθεύσει ότι σε ένα χρόνο έχουν εξασφαλιστεί περαιτέρω πρόοδοι. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κλείνουμε τη συζήτηση αυτή με τον κύριο Ντόρφμαν και μετά θα δώσω αμέσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και πολύ σύντομα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μας δίνεται να γίνει συζήτηση σήμερα και τι μας είπε χθε ε, ο επίτροπο ότι δεν κρίνει το θέμα αυτό ε, δική του αρμοδιότητας αλλά άλλου χαρτοφυλακίου. Θα ήθελα όμως να γνωρίζουμε τι γίνεται ε, Είναι ένα θέμα όμως το οποίο έχει να κάνει και με την ασφάλεια της διατροφής και με τους παραγωγούς μας και γι' αυτό οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει. Θα ήθελα λοιπόν να σημειώσω ότι κάνουμε νομοθεσία, έχουμε εισαγάγει εδώ και χρόνια την νομοθεσία για ασφαλή τρόφιμα για καλά τρόφιμα. Έχουμε ορίσει τις προθεσμίες και τις συνέπειες και δεν είναι δυνατόν ε, μέσα σε ένα περιορισμένο διάστημα να βρεθούν οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί ενώπιον της άρεσης έκπληξης να βρίσκονται αυτοί σε δυσμενές θέσεις από εκείνους που δεν έχουν προσαρμοστεί στην νομοθεσία. Έχω όμως συγκεκριμένε ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ερωτώ μετά την θέση σε εφαρμογή των ε, ε, μεγάλων κλοβών τι θα γίνει με εκείνα τα αυγά τα οποία δεν καταστρέφονται και τα οποία είναι παράνομα. Και επίσης πώς μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για την πράγματι χρήση των νέων αυτών μεγάλων κλοβών. Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται απλώς οι μικροί παλαιοί, οι μικροί κλοβοί να περάσουν τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνεχιστεί εκεί η παραγωγή σε τέτοιου είδου συστοιχίες των αυγών αυτών, τα οποία μετά θα ξαναμπαίνουν ελαθρέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πουληθούν ε, θα, θα ξαναμπαίνουν μάλλον για να πουληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω προϊόντα τρίτων κρατών. Ευχαριστώ. Είναι προφανέ ότι το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο τον κύριο Ντάλι, αλλά και το περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρξει μία λύση στο πρόβλημα αυτό. Ο κύριο Γκαρινέλη έχει το λόγο από την Κομισιόν. Ehm, Ευχαριστώ. Καταρχά, να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γεωργία για την συζήτηση που είχατε και για την ευκαιρία που μου δώσατε να ακούσω αυτό, ζω, ζωντανά αυτό που συχνά μου είχα, είχατε θέσει γραπτό. Λυπάμαι που ορισμένε απαντήσει μου δεν ήταν επαρκώ σαφεί. Στα λίγα λεπτά που έχω στόσο στη διάθεσή μου μπορώ να πω τα εξής δεχόμαστε ευπρόσδεκτα τη συνέχιση της συζήτησης αυτής σε διάφορα επίπεδα και να συνεχίσουμε να αναλύουμε την κατάσταση με ιδιαίτερη προσοχή. Το θέμα για την επισήμανση για της κυκλοφορίας των νομίμων ΟΟΝ ρυθμίζεται σαφώς από κοινοτική νομοθεσία που θα καθαστήσει παράνομη την κυκλοφορία αυγών που εκτρέφονται σε ε, κλοβού που δεν τηρούν τι ε, προδιαγραφέ τη Η Κομισιόν λοιπόν θα φροντίσει ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν ε, την διαδικασία. Η ΔΕΜΗ ξεκινάει η διαδικασία παραπομπή. Ήδη έχουν ξεκινήσει τέτοιε διαδικασίες εναντί κάποιων κρατών μελών με βάση τις εκθέσεις τη Κτηνιατρική Επιτροπή. Πρόκειται για κοινή δράση τόσο νομική όσο και πολιτική. Εγώ μπορώ να σας πω τα στοιχεία. Έγιναν 20 επιθεωρήσεις, 20 έλεγχοι, όλοι είναι διαθέσιμοι οι παρατηρήσει για, για τους τρόπους παρέμβασης με πήγοντα τρόπο για να απαντήσουν στα αιτήματά σα έγιναν. Τα κράτη που παρουσίασαν συγκεκριμένο πρόγραμμα δράση, ωστόσο είναι τέσσερα. Μάλτα, Ρουμανία, Γερμανία, Λιθουανία. Από τα άλλα 25 κράτη-μέλη που επισκέφθηκαμε, παρά το ότι ζητήθηκε να προετοιμάσουν ένα πρόγραμμα παρέμβαση και μια έκθεση για το πώ οι αρμόδιες αρχέ των κρατών μελών θα υλοποιήσουν μία μεταφορά από το ένα σύστημα στο άλλο, δεν απαντήθηκαν. Χωρίς τις απαντήσεις, χωρίς τα στοιχεία αυτά, δεν είναι εύκολο να κάνουμε enforcement. Οι μόνιμες κτηνιατρικές επιτροπές ζήτησαν στοιχεία για τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. Υπάρχει ειδική ε, νομοθετική ρύθμιση που απαιτεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών να δίδουν κάθε χρόνο στοιχεία για ελέγχους και επιθεωρήσεις με τον αριθμό των ε, κοτών που υπάρχουν σε διάφορα συστήματα εκτροφή. Τα στοιχεία αυτά δεν έφτασαν από όλα τα κράτη-μέλη. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίε παραπομπής, είναι διαφανε. διάφανες. Ιδίω κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει την υποχρέωσή του να εφαρμόζουν την νομοθεσία. Όταν λοιπόν έχετε ένα βουλευτή και μιλάει για δυσκολίε εφαρμογή θα πρέπει να δει την δεκαετία αυτή. Τι έγινε η δεκαετία νομοθεσίες για την ευημερία των ζώων στα κράτη-μέλη, που νομοθεσία έδωσε λίγα εργαλεία ελέγχου σε κοινοτικό επίπεδο. Και αυτό είναι από τα βασικά ζητήματα που ανακύπτουν από την αξιολόγηση που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για την πολιτική ευημερία των ζώων. Παρ' όλα αυτά, για να πω και κάτι το θετικό, το σύστημα αγοράς και αυτό που ζητάει η αγορά αλλάζει προς, σαφώς προς τα εναλλακτικά συστήματα που είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ε, σημαντικό ρόλο ποιότητα στην ε, διάσταση εφημερία των ζώων. Τα στοιχεία αυτά έρχονται όχι μόνο στη Γενική Διεύθυνση Καταναλωτών αλλά και στη Γεωργία. Είναι κοινή συζήτηση. Ε, συζήτηση σημαντική όπου θα πρέπει να δώσουμε απάντηση για τα θέματα αναθεώρησης των κοινών ε, πολιτικών. Είναι μια συζήτηση ε, για την οποία ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να έρθουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό σε αυτό το πολύ σημαντικό, σημαντικότερο πλαίσιο έκφραση των πολιτών που είναι το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ε, είναι προφανές από αυτό που μας είπατε ότι πρέπει να συνεχίσουμε την δραστηριότητα ευαισθητοποίηση, διότι προφανώ δεν μπορούμε να σταθούμε αδρανεί. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Άρα θα συνεχίσουμε και στο επίπεδο τη Επιτροπή Γεωργία αλλά και στην Ολομέλεια ζητώντα μια παρέμβαση με προφορική ερώτηση ενδεχομένω. Ο Ζωσέ Μποβέ είναι εδώ ο κύριος Γκαβινέλη και υποφελούμε τη ευκαιρία αυτή ε, γιατί ο κύριος Γκαβινέλη εκπροσωπεί τον κύριο Ντάλι. Για να ενημερώσω τους συναδέλφους στο Κοινοβούλιο ότι σήμερα το πρωί έκανα μια συνέντευξη, έδωσε μια συνέντευξη τύπου για να καταγγείλω την δυσλειτουργία του ΕΦΣΑ και για να καταγγείλω το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΕΦΣΑ εκπροσωπεί σε διεθνές επίπεδο το αγροτικό και το λόμπι το, το, το διατροφικό και ότι στην έκθεση που έδωσε για τις σχέσεις του με τις διάφορες ε, με τους διάφορους κλάδους ε, παραπλάνησε την Επιτροπή τον Μάρτιο όταν το έκανε. Σήμερα η ΕΦΣΑ μετά την ε, μάλλον σήμερα έδωσε τη συνέντευξη, η ΕΦΣΑ άλλαξε τη δήλωση της κυρίας Μπανώτη χτες στις 6 το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν καταγγέλλω το ότι η Επιτροπή καλύπτει, συγκαλύπτει παράνομες δραστηριότητε. Το είπα αυτό, το είχα πει στον κύριο Ντάλη ήδη από τις 14 Ιουλίου. Περίμενα να υπάρξει παρέτηση. Τίποτα. Γι' αυτό τα κοινοποίησα σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση αυτή, θα σας την στείλουμε. Ένα άλλο στοιχείο. Σας στείλαμε το χρονοδιάγραμμα του 11. Εντάξει, δείτε το και θα τα πούμε στις 3. Σε άλλη αίθουσα. Ευχαριστώ.